Dear colleagues, um, I welcome Καλωσορίζω τον οριστή επιτροπό, τον κύριο Julian King, σε αυτή την επιτροπή εσωτερικών υποθέσεων και δομικών ελευθεριών και θα κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις πριν ακούσουμε τις παρατηρήσεις ε, του κύριου Τζουλιαν Κίνγκ και τις ερωτήσεις. Καταρχήν για τη διαδικασία ε, σύμφωνα με το παράρτημα 26 και τις ε, ε, διαδικασίες βάσει των προσωπικής αμεροληψίας και των προσόντων θα εξαρτηθεί θα εξεταστεί και η γνώση του χαρτοφυλακίου του Οριστέντε επιτρέπου. Επίση, έχουμε προετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο για τον Οριστέντε επιτρέπου με δύο κοινέ ερωτήσει που έχουν συνταχθεί από τη Σύνοδο των Προέδρων και τρει ειδικέ ερωτήσει που έχουν προετοιμαστεί από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όλε έχουν επικυρωθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων. Ο επιτρόπο έχει απαντήσει γραπτός και έχουν διανεμηθεί οι απαντήσεις σε όλα τα μέλη, σε όλες τις γλώσσες. Έχετε τις απαντήσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις έχουν και θα ήθελα να τις διαβάσετε αυτές τις απαντήσεις αν δεν το έχετε κάνει ήδη τώρα για τη δομή της συζήτησης οριστής επίτροπος θα κάνει μια εισαγωγική ομιλία για 15 λεπτά. Κατόπιν ε, θα έχουμε 45 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ε, το θα έχουμε χρονοθυρίδα τριών λεπτών, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. Με τη συμφωνία και του κυρίου Μπροκ, μία ερώτηση θα τεθεί από τον κύριο Πάσκου, τον αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ο πρώτο γύρο ρωτήσεων θα τεθεί από του εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων και στο τέλο τη ακρόαση ο οριστής επίτροπο, θα έχει πέντε λεπτά για τελικέ παρατηρήσει. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό ε, στο να γίνει σεβαστό ο χρόνο ομιλία, διαφορετικά δεν θα έχουν χρόνο οι τελευταίοι ομίλητε να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Πρέπει να έχετε πειθαρχία και έτσι θα έχουμε χρόνο στο τέλος για συμπληρωματικές ερωτήσεις. Αν σεβαστείτε το χρόνο υπάρχει αυτή η επιλογή. Η διερμηνία υπάρχει σε 23 γλώσσες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα σας, τη μητρική σας γλώσσα, όμως ε, θα ήθελα να έχετε κατά ότι δεν πρέπει να μιλάτε πολύ γρήγορα. Επίσης, ε, είναι ε, web stream της συνεδρίαση και θα υπάρχει και πρόσβαση σε μια βιντεοσκόπηση αυτής της ακρόασης. Όταν παρακαλώ παίρνετε το λόγο να σηκώνετε και το χέρι σας για να βλέπει και οριστής επιτροπός που βρίσκεστε στην αίθουσα και επίσης για να βοηθήσετε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δύο ακόμη πράγματα έχω να πω πριν να δώσω το λόγο στον Οριστέντε Επίτροπο. Θέλω να αναφέρω δύο σημεία σε σχέση ε, με τη λογοδοσία του και τις ευθύνες του στην επιστολή περιγραφής καθηκόντων ε, που έστειλε ο κ. Γιούκερ στον κύριο Κίνγκ και είπε ότι θα ήθελε να είναι επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας και θα εργαστεί υπό την καθοδήγηση του πρώτου αντιπροέδρου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καλύτερη νομοθεσία, το κράτος δικαίου και το η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα υποστηριχθεί και από τον Αρμόδιο Επίτροπο για τη μετανάστευση και τα εσωτερικά θέματα. Επίσης, ο Επίτροπος ε, Μετανάστευσης Ιστορικών Υποθέσεων θα τον βοηθήσει σε οκτώ συγκεκριμένα καθήκοντα. Θέλουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, του κυρίου Κίνγκ και πώς θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους επιτρόπους. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τις γραμμές λογοδοσίας σε αυτή την ακρόαση. Επίσης, διαβάσαμε ότι η προσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επί του Συμβουλίου για θέματα που έχουν να κάνουν με την Ένωση Ασφάλειας ως κανόνας θα διασφαλίζει από την Επίτροπο Μετανάστευση Εσωτερικών Υποθέσεων και Θαγένεια, εκτό αν αποφασιστεί διαφορετικά, αναπερίπτωση από τον πρώτο αντιπρόεδρο. Σε συμφωνία με τον Επίτροπο για την Μετανάστευση και τι Εσωτερικές υποθέσει. σίγουρα κ. Τζούλιαν Κίνγκ θα μα διαφωτίσει πώ θα γίνει αυτό στην πράξη, έτσι ώστε να διασκεδάσει δεξιφώς εδώ σε αυτή την Επιτροπή σε αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ σημαντική η λογοδοσία του σε αυτή την επιτροπή και σίγουρα θα συμφωνεί. Ξέρω ότι ο κ. Τζουλίν Κίνγκ έχει στείλει και γραπτέ απαντήσει και μαζί με την επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα έχουμε επικοδομητικό διάλογο για να δούμε ποιε θα είναι οι προτεραιότητε ε, και πώς θα υπάρξουν αποτελέσματα με πιο διαρθρωμένο τρόπο των θεμάτων που θα έχουν συζητηθεί. Έτσι λοιπόν αυτά τα κύρια θέματα της ευθύνη και της λογοδοσίας για αυτή την Επιτροπή θα ήθελα να φέρω και τώρα θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο στον Εριστέντα Επίτροπο για την παρουσίασή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή ακρόαση. Αν μου έλεγε κάποιο πριν από λίγου μήνε ότι θα ήμουν εδώ ενώπιον σα, ε, δεν θα τον είχα πιστέψει. Βιώνουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Έχω την τιμή να διοριστώ ω υποψήφιο επίτροπο από την Βρετανική κυβέρνηση. Ο πρόεδρο Γιούνκερ έδραξε, την ευκαιρία για να ενισχύσει την Επιτροπή, δημιουργώντας αυτή τη νέα θέση Επίτροπος αρμόδιο για θέματα ασφάλειας. Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν, μα ένας Επίτροπος που διορίζεται από ένα κράτος μέλος που είχε αποφασίσει όμως να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς γίνεται να ε, ε, ε, επιτελέσει ένα ρόλο τόσο σημαντικό. Σας διαβεβαιώ όμως μπορώ να προσφέρω προστιθέμενη αξία σε αυτό το τομέα που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους πολίτες. Έχω συγκεκριμένη εμπειρία στον τομέα αυτό με την ε, από τις θέσεις που κατήχα στο Συμβούλιο αλλά και επιτόπου στην Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία και πιο πρόσφατα στο Παρίσι. Πριν από δύο μήνες ήμουνα στην Ίκαια στις 15 Ιουλίου το πρωί και η διεισόμαση διαπίστωσα ποιες είναι οι καταστροφικές επιπτώσεις της επίθεσης που είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ. Με τόσα θύματα, τόσους τραυματίες που ε, ήταν μια τραυματική εμπειρία για ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλη μια φορά ε, συνειδητοποίησα ποιο είναι το πελώριο ανθρώπινο κόστος της τρομοκρατίας. Αφιέρωσα τη ζωή μου στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, σε διάφορες θέσεις στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο αλλά και στην Επιτροπή. Ήμουν επικεφαλής του Γραφείου Δύο Επιτρόπων. Ήμουν πρέσβης στη Γαλλία και ε, υπερασπίστηκα στεναρά τη θέση της Βρετανικής κυβέρνησης ε, κατά την προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα. Εγώ ανέκαθεν ήμουν περήφανος ε, για την υπηκότητά μου και ταυτόχρονα πολύ περήφανος που είμαι Ευρωπαίος. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίφαση ανάμεσα στα δύο. Στις 23 Ιουνίου όμως η πλειοψηφία των συμπατριωτών μου αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οφείλουμε να σεβαστούμε την αποφασή τους. Για να διασκεδάσω κάθε αμφιβολία θέλω να ε, με απόλυτη σαφήνεια να αναφέρω ότι αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτελέσω τα καθήκοντά μου περασπίζοντας το κοινό ευρωπαϊκό καλό και μόνο αυτό. Έχω πλήρη επίγνωση του επίπεδου αικαιρεότητας, αμεροληψίας και ευρωπαϊκής δέσμευσης που περιμένετε προσδοκάτε ε, θεμητά από μένα εάν μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας ε, διοριστός επίτροπος ε, θα επομισθώ όλες αυτές που επισύρει αυτός ο διορισμός. Έχουν περάσει 15 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Πώς ε, σκεφτόμαστε απέναντι σε τέτοιες απειλές και πώς αντιδρούμε έχει αλλάξει. Αλλά τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα εξακολουθούν να απειλούν τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας. Και κάποιοι θα έλεγαν σήμερα περισσότερο από ποτέ από τους βομβαρδισμούς της Μαδρίτης το 2004 είχαμε δεκάδες ε, άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις. 14 μόνο πέρσι με 600 άτομα τα οποία σκοτώθηκαν. Κάποιες από αυτές τις επιθέσεις ήταν πολύ προγραμματισμένες από ομάδες, άλλες ήταν επιθέσεις ε, με ένα μαχαίρι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ε, τρομοκράτες είχαν μεγαλώσει εδώ, άλλοι όμως είχαν επιστρέψει από το εξωτερικό που είχαν πολεμήσει. Κάποιοι ήταν υπό παρακολούθηση, άλλοι ήταν γνωστοί στις αρχές ε, και είχαν ποινικό μητρό για μικρό εγκλήματα. Κάποιοι ήταν ε, πολύ πιο κοντά στους δρομοκράτες, άλλοι ριζοσπαστικοποιήθηκαν σε ένα διάστημα εβδομάδων. Κάποιες επιθέσεις έγιναν σε ευαίσθητους στόχους, άλλες ήταν τελείως ε, αναπάντεχες και βεβαίως στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος αναπτύσσονται νέοι τρόποι το κυβερνοέγκλημα αναπτύσσεται καθημερινά και γίνεται όλο και πιο επιθετικό και απειλεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και την οικονομία. Ούτε η τρομοκρατία, ούτε το οργανωμένο έγκλημα σέβονται τα εθνικά σύνορα. Μάλιστα, έτσι ακριβώ λειτουργούν από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ κρατών. Υπάρχει προφανώ, μια ευρωπαϊκή διάσταση. Δείτε τι επιθέσει στο Παρίσι τον Νοέμβριο που μα πέρασε. Σχεδιάστηκαν στη Συρία. Κάποιοι από του τρομοκράτε, από ό,τι φαίνεται ταξίδευσαν με ψεύτικα διαβατήρια. Μετά έμειναν στο Βέλγιο όπου βρήκαν όπλα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια και πήγαν στη Γαλλία την προηγουμένη τη επιθέσεω μόνο. Δεδομένων λοιπόν αυτών των πολυεθνικών εφοδιαστικών αλυσίδων, ο μόνο τρόπο να νικήσουμε του τρομοκράτε και του εγκληματίε είναι μέσω τη αποτελεσματική συνεργασία. Στον σημερινό κόσμο η ασφάλεια του ενό κρατου μέλου είναι η ασφάλεια όλων μα. Και βέβαια στο άρθρο 4 τη συνθήκη είναι σαφέ. Η εθνική ασφάλεια παραμένει αρμοδιότητα αποκλειστική των κρατών μελών. Αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο του απειλέ, οι οποίε είναι διεθνεί. Γι' αυτό ακριβώ χρειάζεται αυτή η θέση αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι αυξανόμενε απειλέ απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας αφαιρέσουν την ελευθερία μας και τα θεμελιώδη δικαιώματα, πράγματα για τα οποία έχουμε παλέψει σκληρά. Επίσης, είναι αυτό το οποίο περιμένουν οι πολίτες μας. Το Ευρωπαρόμετρο βρήκε πως 82% των όσων απάντησαν ζήτησαν ισχυρότερη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αντιδρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά εντό της Κομισιόν με τον πρώτο αντιπρόεδρο τον κύριο Τίμερμανς, τον κύριο Βραμόπουλο, την κυρία Γιούροβα και όλους τους άλλους συναδέλφους επιτρόπους. Σε αυτό το πνεύμα, όπως αναφέρεται εξάλλου και στην επιστολή που μου απίφθινε ο πρόεδρος Γιούνκερ, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας οριζόντια με προσωπικό από τις διάφορες διευθύνσεις της Κομισιόν την Διεύθυνση Δικαιοσύνη, Εσωτερικών Μεταφορών και Εκπαίδευση. Επίση, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμό και κοινή εργασία με τα κράτη-μέλη και με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σα. Γνωρίζω πώ εσεί θέλετε ακριβώ να πετύχει το θέμα τη ασφάλεια και την ενέργεια την οποία αφιερώνεται για να σημειωθεί πρόοδο σε πολλέ προτάσει. Πρέπει λοιπόν τώρα να αυξήσουμε τι προσπαθίε μα για να μπορέσουμε να παρέχουμε την ασφάλεια που θέλουν οι πολίτες μας. Πρέπει να υπάρξει μια αποτελεσματική και βιώσιμη ένωση ασφαλείας. Αποτελεσματική σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάζουμε συνεχώς στην εφαρμογή. Να μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο τα συμπεφωνημένα, να βοηθάμε τις εθνικές αρχές να δουν ποια είναι τα εμπόδια στην εφαρμογή και να τα αντιμετωπίζουμε μαζί και βεβαίως τα εφιστάμενα συστήματα να χρησιμοποιούνται πλήρως. Τα κράτη-μέλη μπορούν να βασίζονται στην Κομισιόν για βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όταν αυτό είναι αναγκαίο δεν θα διστάσουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο και χρησιμοποιώντας διαδικασίες επί παραβάση. Αλλά βεβαίως ας πρέπει πρώτα απ' όλα να εργαστούμε στον τομέα της εφαρμογής. Βιώσιμη Ένωση Ασφάλειας συνεχείς αυτές τις επιθέσεις σημαίνουν πως δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια συνολική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να είναι διαρκής σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφαλείας. Και βεβαίω τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να είναι στην καρδιά αυτού του πλαισίου. Η δική μου εμπειρία στη Βόρεια Ιρλανδία με έχει διδάξει πω η ειρήνη και η μεγαλύτερη άρα ασφάλεια μπορεί να υλοποιηθεί μόνο όταν βασίζεται στον πλήρη σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας στην Βόρεια Ιρλανδία σημείωσε πρόοδο όταν οι άνθρωποι πίστευσαν ότι τα θεμελιώδη τους δικαιώματα θα γινόταν σεβαστά και έτσι μπόρεσαν να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον. Είμαι λοιπόν απολύτω προσιλωμένο στον χάρτη. Οι δράσει μα θα πρέπει πάντα να βασίζονται στο κράτο δικαίου με τι απαρότητε ε, δικλείδε ασφαλεία και εξαιρέσει μόνο όταν είναι αυτό αναγκαίο, αναλογικό και αιτιολογείται νομικά. Όσον αφορά τι προτεραιότητε μου, η φετηρία είναι η ανακοίνωση τη Κομισιόν του Απριλίου 2016 για μια, ασφάλεια, για μια ένωση ασφαλεία. Και έτσι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τον κοινό μα αγώνα κατά της τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τι άμυνές μα απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και την αντοχή μα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να συμφωνήσουμε επιγόντω επί της πρότασης για μια οδηγία καταπολέμησης τρομοκρατίας. Σε συνεργασία με εσά και το Συμβούλιο ελπίζω αυτό να γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης πρέπει να κόψουμε την πρόσβαση των τρομοκρατών σε χρηματοδότηση. Η Κομισιόν θα καταθέσει τις σχετικές προτάσεις για τα πυροβολά όπλα. Για εμένα μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μειωθεί η πρόσβαση στα παράνομα όπλα. Πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή του σχεδίου δράσης Και εδώ πέρα, όπω και αλλού, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Δεύτερον, οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικότερο ρόλο για να στηρίξουν τις εθνικές αρχές προσπάθειές τους κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ πάντα θα υπερασπίζομαι την Europol. Τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες που μας προσφέρει το νέο νομικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας της Europol έχει αρχίσει να λειτουργεί, αλλά πρέπει να το ενισχύσουμε και άλλο. Επίσης, Πρέπει να στηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματο, έτσι ώστε να γίνει ο κύριος κατά καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματο και να λάβει υπόψη την τρομοκρατική απειλή. Οι υπηρεσίε επιβολή του νόμου, τα σώματα ασφαλεία θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ερευνούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά στοιχεία και οι εθνικέ αρχέ θα πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο τι κοινέ ομάδε έρευνα με τη βοήθεια τη Europol και του Eurojust. Τρίτον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ριζοσπαστικοποίηση που μπορεί να οδηγήσει σε βίαιο εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στα παιδιά και τους νέους. Έχουμε λοιπόν το δίκτυο ενημέρωσης για την ριζοσπαστικοποίηση που βασίζεται σε μια προσέγγιση συνεργατική και έχει ήδη αποτελέσματα βοηθώντας όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στις φυλακές και στα σχολεία. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να στηρίξουμε και την κοινωνία των πολιτών για να αναπτύξει κάποια άλλα αφηγήματα. Τέταρτον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα των τρομοκρατών και την προπαγάνδα του μίσου στο διαδίκτυο. Πέρα από αυτά τα οποία σας ανέφερα, πρέπει να δούμε την δυνατότητα μιας κοινή πλατφόρμας καταγγελιών με τον κλάδο για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείε των ε, κοινωνικών μέσων για να κατεβάζουν απαράδεκτο περιεχόμενο. Όπως είπα, πρέπει να ενισχύσουμε τις άμυνές μας απέναντι στην τρομοκρατία, να ενισχύσουμε την αντοχή μας και να βελτιώσουμε περισσότερο το πώς συνεργαζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες. Οπότε πέμπτον, τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Παραδείγματος χάρη δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση του ΠΡΟΜ. Αντιμετωπίζουμε επίσης σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος ε, της οδηγίας για τα στοιχεία αεροπορικών επιβατών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν το σύστημα να λειτουργήσει. Έκτον, πέρα από τα εφιστάμενα συστήματα τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν, πρέπει να δούμε πώς μοιραζόμαστε πληροφορίες μεταξύ των συστημάτων μας. Τα εφιστάμενα συστήματα είναι περίπλοκα και κατακαιρματισμένα. Σεβόμενοι του περιορισμού πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τι πληροφορίε στο επίπεδο τη Ένωση. Πρέπει επίση να έχουμε ποιοτικά δεδομένα να υπάρχει η κατάλληλη επεξεργασία και να είναι διαθέσιμα στους κατάλληλους ανθρώπους όταν τα χρειάζονται, πάντα σεβόμενοι τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσω της ομάδας υψηλού επίπεδου για τα συστήματα πληροφορικής. Έβδομον, πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα. Οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες δρούν διασυνοριακά και η έλεγχη στα εξωτερικά σύνορα είναι ένας τρόπος κλειδί για να τους σταματήσουμε το προτινόμενο σύστημα εισόδου-εξόδου είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώ θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων. Ε, το προτινόμενο σύστημα ETIAS για την πρώτερη αδειοδότηση σημαίνει ότι θα έχουμε και πρώτερους ελέγχους ασφαλείας για επικόους τρίτων χωρών και η Ευρωπαϊκή Συνορία Φιλελεακή και Ακτοφυλακή θα αρχίσει να επιχειρεί σύντομα. Επίσης, η έλεγχοι στα σύνορα θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο, και τα δίκτυα λάθροδιακίνησης, καθώς επίσης και να ταυτοποιήσουμε όσους επιστρέφουν ενώ είχαν πάει να πολεμήσουν στο εξωτερικό. Αλλά δεν ναι, θα πρέπει να μπερδεύουμε τα ζητήματα της τρομοκρατίας με τα ζητήματα μετανάστευσης ή ταυτότητας. Έτσι θα ενισχύσουμε, αν το κάνουμε αυτό, θα ενισχύσουμε τον λαϊκισμό ο οποίος στιγματίζει ευάλωτους πληθυσμούς. Όγδον, πρέπει να ενισχύσουμε την δυνατότητά μας να προστατεύσουμε κρίσιμες υποδομές και εύκολους στόχους. Οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν δείξει πού είναι οι αδυναμίες. Η έρευνα και οι νέε τεχνολογίε μπορούν να βοηθήσουν. Η σημαντική η πρόοδο έχει γίνει στον τομέα τη ασφαλή αεροπορία. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και στην ασφάλεια στην ε, θάλασσα και βεβαίω στην κυβερνοασφάλεια. Τέλο, πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με τα θύματα τη τρομοκρατία. Είχαμε περάσει την πρόσφατη αναθεώρηση τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά στο μέλλον. Θα ήθελα να καταλήξω λέγοντα λίγα λόγια για το πώ θεωρώ ότι θα συνεργαστώ μαζί σα στην ε, ΛΥΜΠΕ. Πέρα από συνομοθέτη, είστε επίση μια πηγή ιδεών και έμπνευση. Μπορείτε να ασκήσετε πολιτική πίεση έτσι ώστε να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα και να μας βοηθήσετε με τα αποτελέσματα και την εφαρμογή. Πιστεύω πως θα πρέπει το εκτελεστικό, η εκτελεστική εξουσία να είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο. Και πέρα από οποιαδήποτε επίσημη δική σας πρόσκληση, ευχαρίστως θα ε, έρχομαι εδώ πέρα για να σας λέω ότι γίνεται σε τακτική βάση. Έχετε ζητήσει πολλές φορές, για μια, έχετε ζητήσει πολλές φορές μια πιο συνολική επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων πολιτικών μας κατά της τρομοκρατίας. Συμφωνώ και θέλω να συνεργαστώ μαζί σας. Επίσης, πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε περισσότερη επιχειρησιακή γνώση λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη φύση αυτών των πληροφοριών. Θέλω λοιπόν να συνεργαστώ μαζί σας για να προχωρήσουν αυτά τα ζητήματα. Εάν λοιπόν με επιβεβαιώσετε στη θέση αυτή, θα εργαστώ άοκνα με εσάς, με τους συναδέλφους μου στην Κομισιόν, για να κλείσουμε τον χώρο στον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επιτεθούν σε ελευθερίες μας για να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ασφαλή για τους πολίτες με περισσότερη συμπερίληψη για όλους και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Αυτό θα γίνει πάντα με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία θέλουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε γιατί χωρίς αυτά θα έχουμε αποτύχει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Κύριε Ρεστέντε και τώρα περνάμε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων που θα γίνει από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα ξεκινήσουμε με το, τη συντονίστρια του ΕΛ, το συντονιστή του ΕΛ, Ρομπέρτο Μετσούλα. Ένα λεπτό για την ερώτηση. Ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας εδώ απόψε και για την ανακτήρια δηλωσή σας. Καθώς ε, είμαι πρώτη που θέτω ερώτηση, θα μπορείτε να πείτε κάποιες ε, περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι θα κάνετε για να προωθήσετε μια ένωση ασφάλεια στο δύσκολο κλίμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη και ιδίω ε, εφόσον έχουμε συνεχείς διακυβερνητικές προσεγγίσεις για θέματα ασφάλειας και ποιες προσπάθειες θα κάνετε έχοντας κατά νου τις αντίστοιχες αρμοδιότητες αλλά κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς μαχητές για να ε, προωθήσετε την ανάκληση των διαβατηρίων. Θα διερευνήσετε κάτι τέτοιο ως πιθανό μέτρο για το πώς θα αντιμετωπίσετε τις σύγχρονες απειλές που έχουμε με τους ξένους μαχητές που έχουν διπλή υπηκότητα. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Μπόρεσα να σας εντοπίσω, αλλά είναι μεγάλη αίθουσα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ε, σας ζητήσω την ανεκτικότητά σας αν ψάχνω να εντοπίσω κάποιον στην αίθουσα. Συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε για την ε, ανάγκη για μια πλήρη και συντονισμένη και σε πολλαπλό επίπεδα απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά δρούμε στο πλαίσιο των συνθήκων, αλλά ε, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνο τους. Νομίζω έχει σαφή ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Πολλά μπορούμε να συνεισφέρουμε. Μπορούμε να συνεισφέρουμε τους οργανισμούς μας, τα συστήματά μας, τα συστήματα πληροφοριών και άλλα. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην ενίσχυση των συνόρων, αλλά και πίσω από τα σύνορα με την με την ορθή χρήση του ΣΥΣ μπορούμε να παρουσιάσουμε νομοθεσία που θα θέσει πρότυπα, όπω παραδείγματο χάρη για την καταπολέμηση τη νομοποίησης παράνομων εσόδων ε, και σκέφτομαι παραδείγματο χάρη την ενίσχυση τη συνεργασία, όπω ε, ε, το ένταλμα έρευνα, που θα έρθει την Άνοιξη και μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο. Ανέφερα το εξαιρετικό δίκτυο για την ευαισθητοποίηση, για την ριζοσπαστικοποίηση. Μπορούμε να δώσουμε χρηματοδότηση φυσικά και του ISF και μέσω του ορίζοντα 2020 και συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σειρά πραγμάτων να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα για τη συγκεκριμένη ερώτηση που θέσατε για τα διαβατήρια και για τους ξένους μαχητές. Τώρα το θέμα φυσικά ε, των διαβατηρίων αλλά και τη υπηκότητα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να λάβουν δράση για τα διαβατήρια και φυσικά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αρνηθούν την είσοδο ή να απελάσουν κάποιον για λόγους δημοσίας ασφάλειας. Έτσι λοιπόν αυτό είναι κάτι που θα ήθελα ε, να το συνεχίσω, να δώσω συνέχεια συνεργασία με την κυρία Γιούροβε. Τώρα, η κυρία Σίπελ από το SND. Ευχαριστώ. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει καλέσει εδώ και καιρό για πλήρη αναθεώρηση των φυστάμενων μέτρων Τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα για να αξιολογήσουμε τι δουλεύει σωστά, που είναι οι ελλείψεις και τα κενά στην εφαρμογή. Στο ρόλο σας ως Επίτροπο για την Ένωση Ασφάλειας ε, θα κάνετε μια τέτοια αξιολόγηση κυρίως σε ό,τι αφορά την ε, ενασχόλησή σας να βρείτε τις ελλείψεις και να τις καλύψετε και να καλύψετε τα κενά και πώς θα προχωρήσετε σε αυτό το θέμα. Και έχω και μια δεύτερη ερώτηση για να επερασπίσουμε τις ελεύθερες και δημοκρατικές κοινωνίες μας. Πώς θα εγγυηθείτε ότι όλα τα μέτρα που προτείνονται από την Κομισιόν σέβονται τις αρχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κυρίως την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Ευχαριστώ. Όπως είπα στο τέλος των παρατηρήσεών μου, συμφωνώ με όσους ζητήσατε αναθεώρηση των ε, σημερινών πολιτικών στον τομέα. Αν με επιβεβαιώσετε, ο διορισμός μου σε αυτό το ρόλο θα συνδράμει σε αυτό φυσικά. Ε, κάποιοι αντιτίθεται ε, στον ελευθερή δραστηριότητα. Εγώ νομίζω ότι αν συνεργαστούμε μαζί για να βρούμε τους συγκεκριμένους τρόπους θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αναθεώρηση και μια αναθεώρηση γιατί το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για το ποιο αντίκτυπο έχει αυτό στα κράτη-μέλη και εντό των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν κάνω αυτή τη δέσμευση απέναντί σας για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, που φυσικά είναι κρίσιμο σημείο όλου του πλαισίου στο οποίο εργαζόμαστε, θα ήθελα να είμαι πολύ το σαφής. Εδώ εμείς έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο έχει προσδιοριστεί από ορισμένε αποφάσεις πολύ διάσημες και βλέπετε ότι τώρα υπάρχουν σε διάφορες γνωμοδοτήσεις. Εγώ δέχομαι αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το σωστό πλαίσιο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε μια βιώσιμη ένωση ασφάλειας. Όπως είπατε, θα πρέπει οι εξαιρέσεις να είναι αναγκαίες, αναλογικές και νόμιμες. Έχουμε αυστηρούς κανόνες για τη χρήση και για την πρόσβαση και θα πρέπει να σεβαστούμε ε, και και τους ε, περιορισμούς σε σχέση με το σκοπό και τη διάρκεια. Ευχαριστώ. Από το συντονιστή του ΕΣΥΑΡ, τον κύριο Κυρκόπα, είναι η τρίτη ερώτηση. Τζούλιαν, μπορείς ε, να διαβεβαιώσεις στα μέλη αυτής της Επιτροπής ότι η Ένωση Ασφαλείας ε, δεν θα ξεπεράσει τις αρμοδιότητές της και θα διατηρήσει σαφή διαχωρισμό μεταξύ της ε, εθνικής συλλογής πληροφοριών και της ανταλλαγής πληροφοριών ε, σε διασυνοριακό επίπεδο και πώς βλέπεις ότι θα αναπτυχθεί ε, αυτός ο τομέας στα επόμενα χρόνια κυρίως αν υπάρξει υπέρβαση από αυτό που προβλέπουν οι συνθήκες και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξή. Εγώ ήμουν εισηγητή για τι κοινέ ερευνητικέ ομάδε το 2001. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιε μεικτέ απόψει για την επιτυχία των ομάδων αυτών. Ε, θα παρουσιάσει μία αναφερμένη πρόταση για τι κοινέ ερευνητικέ ομάδε, καθώ υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία στις αντιδρομοκρατικές έρευνες. Ευχαριστώ. Όπως είπα, όταν απαντήσα την πρώτη ερώτηση, είμαι σαφής στο ότι λειτουργούμε εντός του πλαισίου των συνθήκων. Λεχθέντος αυτού, νομίζω ότι πολλά μπορούμε και θα έπρεπε να κάνουμε εντός αυτού του πλαισίου. Αυτές οι απειλές που αντιμετωπίζουμε και που έχω περιγράψει, εν συντομία, είναι κοινέ απειλέ και μας φύγουν όλους σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια και θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να απαντήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, γιατί τα συστήματα δεν θα λειτουργήσουν αν οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται. Νομίζω ότι έχουμε εδώ μία ευκαιρία τώρα και αυτό σχετίζεται με την ερώτησή σας, με την ε, ε, ενίσχυση της Europol και ε, την δημιουργία του ECTC, του κέντρου, για να μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτού του είδους την εμπιστοσύνη με τα κράτη-μέλη και με τις διάφορες εθνικές αρχές. Και μετά τις επιθέσεις του Παρισιού, η συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και των Βελγικών και των Γαλλικών αρχών θα γνωρίζετε την επιχείρηση αυτή. Αυτό το παράδειγμα μου δίνει την εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια τέτοια πρακτική και σταθερή συνεργασία. Πολλά μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια των συνθήκων για τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Υποστηρίζω την ιδέα ότι θα πρέπει να κάνουμε πολλά για να ενθαρρύνουμε τις εθνικές αρχές να εκμεταλλευτούν τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες και με κάπως μιλώντας με ανθρώπους που έχουν εργαστεί σε αυτό το τομέα πρόσφατα που κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει τόσο όσο θα περιμέναμε. Και πάλι ελπίζω ότι τα θετικά παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας όπως ε, οι επιχείρησεις φροντιτεχνητέ θα ενθαρρύνουν τη χρήση τέτοιων κοινωνικών ομάδων όχι μόνο με τη Europol αλλά και με τη Eurojust και θα μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και με άλλους οργανισμούς και με τις συνοριοφύλακες από την συντονίστρια του κυρία Βίξτρομ, παρακαλώ, θα κάνει την δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διευθύντε Επίτροπε, θα ήθελα από πλευρά των Φιλελευθέρων να σας καλωσορίσω. Σας έχει ανατεθεί ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο Δυστυχώς ε, υπάρχει κατάχρηση από κάποιους που θέλουν να διαιρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε- Ένωση της Ασφάλειας είναι κάτι που πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες. Πώς μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε τις επικείμενες ε, συζητήσεις για τα θέματα ασφάλειας. Θα βασιζόμαστε σε τεκμήρια, σε γεγονότα, ή σε συγκεκριμένα στοιχεία και μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει μια σαφής διάκριση αφενός ανάμεσα στην πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωση και αφετέρου ανάμεσα στη μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου. Και επίσης ε, ενώ διάφορα εργαλεία για την ασφάλεια εφαρμόζονται τώρα η πρόληψη της ρουσπαστικοποίησης ε, και του βίαιου εξτρεμισμού φαίνεται να υστερούν. Πολύ συγκεκριμένα, ποιες είναι οι συστάσεις σας για να επιταχύνουμε, να εντετικοποιήσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε σε αυτό το τομέα. Προκρίνεται μια ανεξισορρόπηση των μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ε, ριζοσπαστικοποίηση και του βίου εξτρεμισμού, κυρίως σε επίπεδο τοπικών αρχών και την ε, καταπολέμηση του ρατσισμού και της στιγματοποίησης ε, συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων. Απάντηση. Ευχαριστώ, όπως είπα, στις μου παρατηρήσεις. Ε, ο μόνος τρόπος και δρόμος που γνωρίζω εγώ για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές μας είναι να βασιζόμαστε σε τεκμήρια, σε αποδείξεις. Κατά παράδοση έτσι λειτουργώ και έχω την πρόθεση να συνεχίσω έτσι. Ο μηχανισμός, ακριβής μηχανισμός που, ε, τον οποίο θα ακολουθήσουμε σε διάφορες αρχές είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Είτε μιλάμε για την πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών ε, ε, είτε πρόκειται για την συγκρότηση του ίδιου του μηχανισμού, αυτά θα τα συζητήσουμε ε, στην πορεία. Όμως σίγουρα θα βασιστούμε σε συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια για τη μετανάστευση. Όπω σα είπα και στι ε, προκατοικές μου παρατηρήσει, φυσικά πρέπει να υπάρχει σαφή διάκριση ανάμεσα στι δύο πολιτικέ ασφάλεια, Αφενό και μετανάστευση και ασύλου αφετέρου. Ε, χαιρετίζω την δράση του Επίτροπου Αβραμόπουλου για, στον τομέα τη μετανάστευση Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνουμε εμεί ε, στον τομέα τη ασφάλεια. Υπάρχουν κάποια περιστατικά ε, όπου χρησιμοποιούν μεταναστευτικέ οδού ε, οι τρομοκράτε ε, για να επανέλθουν αυτά φτάσουν στην Ευρώπη και γι' αυτό είναι σημαντικό και έχουμε κάνει σχετικά βήματα και τα θέλαμε να ενισχύσουμε τα hot spots και να επεκταθούν αυτές οι βέλτιστες πρακτικές και οι πρακτικές ρυθμίσεις που έχουμε στα σύνορά μας αλλά σίγουρα θα πρέπει να ε, ε, εφαρμόζουμε τις αρχές μας για θεμελιώδει θεμελιώδεις ελευθερίες και φυσικά θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις δύο πολιτικές όπως σωστά είπατε. Τρίτο σκέλος ε, για την πρόληψη της ρουσπαστικοποίησης. Ε, σε πολύ διαφορετικές περιστάσεις έχω βιώσει κάτι αντίστοιχο στην Βόρεια Ιρλανδία και από την προσωπική μου εμπειρία θα έλεγα είναι κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε ε, αν δεν συμμετέχετε επί τόπου. Δεν γίνεται παρά να συνεργαστούμε με ε, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με τοπικές αρχές. Το δίκτυο ΡΑΝ, χαίρομαι πάρα πολύ, λειτουργεί και ακριβώς βασίζεται σε αυτά τα ε, δίκτυα τοπικών ε, φορέων και ό,τι μπορώ να κάνω για να υποστηρίξω τις προασπού τους στην Ευρώπη θα το κάνω με μεγάλη χαρά. Ερώτηση 5 από την ε, Κορνίλια Ένστα. Ναι, εδώ είμαι. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα να μάθω πώς θα διαχωρίσετε τη δικιά σας τη δουλειά από αυτή του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν έχετε δική σας γενική διεύθυνση. Ποιος θα σας συμβουλεύει, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Δεύτερον, με αυτά τα, έχει σχέση με αυτά τα οποία μας είπατε. Θέλετε να εφαρμόσετε τους νόμους, αλλά βεβαίω τίθεται και το ζήτημα της συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τι θα κάνετε όμως εάν ε, το δικαστήριο ακολουθήσει αυτά τα οποία πρότεινε ο εισαγγελέα για τη σύμβαση ε, δεδομένων αεροπορικών υπηρετών με τον Καναδά και την απορρίψη. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Thank you. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση γιατί αφορά τα πρακτικά της συνεργασίας μας. Και πάλι είναι θέμα της νοοτροπίας μου. Εγώ είμαι μαθημένος σε μια νοοτροπία συνεργασίας, σε ομάδες, οπότε είναι τελείως φυσικό για εμένα η βασική επιτροπή στον τομέα αυτών να συνεργάζονται σαν ομάδα. Και τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει από τους πολίτες μας έτοιμα, ε, έντονο μάλιστα, για ε, κινητοποίηση σε αυτόν τον τομέα, εγώ θα θεωρούσα εαυτόν ε, έναν επιπλέον πόρο για να βοηθήσω και εσάς για να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες μας. Και δεν είναι μόνο με τον Επιτροπό Αβραμόπουλο που θα συνεργαστώ. Αν δούμε παραδείγματος χάρη το τι πρέπει να γίνει στον τομέα της ριζοσπαστικοποίηση, σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, δούμε το θέμα αυτό με την νεολαία, την εκπαίδευση, την οικονομική στήριξη. Και θα ήθελα εγώ να συνεργαστώ με πολλούς ε, συναδέλφους. Γι' αυτό είναι θετικό το ότι ο πρόεδρος δημιούργησε αυτή την ομάδα εργασίας. Την τελευταία φορά που ήμουν στην Κομισιόν ήμουν σε μια γενική διεύθυνση την οποία δεν θα κατονομάσω, αλλά δούλευε απομονωμένη. Μια φορά αυτό λειτουργούσε, άλλες φορές όχι. Οπότε είμαι υπέρ αυτής της ομάδας εργασίας η οποία θα είναι οριζόντια εντός της ε, Κομισιόν. Για το ευρωπαϊκό δίκαιο, τον σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου, οπωσδήποτε Είμαι προσιλωμένο σε αυτό. Αναφέρατε την ε, συμφωνία με τον Καναδά. Προφανώς έχω διαβάσει τα όσα προτείνει ο Γενικό. Ε, ο Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η απόφαση τελικά του δικαστηρίου και ε, θα γίνει σεβαστή. Question number for the Greens. Ερώτηση 6 για ε, τους πράσινους, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Κύριε Κίνγκ, Είπατε ότι θα πρέπει να αναχαιτήσουμε την πρόσβαση των προκρατών στη χρηματοδότηση και επειδή εγώ ασχολούμαι με την οδηγία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ήθελα να σχολιάσω το ζήτημα των καταπιστευμάτων που χρησιμοποιούνται από τους τρομοκράτες για τη χρηματοδότηση. Τέτοια τρας ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες. Ε, και επειδή είστε Βρετανός, ε, τι έχετε να πείτε για τα βρετανικά τρας και μπορούμε να υποστηρίζουμε στη βοήθεια σας ε, για να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα των τρας. Δεύτερο ερώτημα. Έχετε μακρά σταδιοδρομία ως δημόσιος υπάλληλος. Πολιτική όμως εμπειρία δεν έχετε καταδείξει. Όχι ότι αμφιβάλλω τις ικανότητές σας. Θέλω να καταλάβω όμως γιατί η Βρετανική κυβέρνηση δεν διόρισε ένα πολιτικό πρόσωπο πρόσωπο σε αυτή τη θέση. Θέλει να αποπολιτικοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Βρετανική κυβέρνηση και θέλει τι διαπραγματεύσει για το Brexit να τι κάνει ε, ε εν πωλής ή και αποκλειστικά μόνο με το Συμβούλιο. Να το ερμηνεύσω έτσι. Ευχαριστώ. Να αρχίσω από το τέλο. αν μου επιτρέπετε. Δεν είμαι πολιτικός, όμως τα τελευταία 25 χρόνια ε, κολυμπώ σε έναν ωκεανό πολιτικό. Ε, και ε, πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα μπορώ να χρησιμοποιήσω τις πολιτικές δεξιότητες που έχω αποκτήσει για να προωθήσω τα ζητήματα. Δεν θεωρώ ότι ο ρόλος αυτός ε, είναι υποδεέστερος. Εγώ ε, σέβομαι την εμπιστοσύνη του Πρόεδρου Γιούγκερ και θα ε, εργαστώ πάρα πολύ σκληρά για να προωθήσω αυτά τα θέματα και να του ξεπληρώσω αυτή τη τιμή που μου κάνει. Ο ρόλος μου σε αυτόν τον τομέα ή σε σχέση με το γενικότερο ζήτημα του Brexit ε, πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν είμαι εκπρόσωπος εδώ της Βρετανικής κυβέρνησης. Εάν θέλουν κάποιοι να κάνουν ερωτήσεις για το Brexit ή για τη θέση της Βρετανικής κυβέρνησης για αυτό το ζήτημα, φοβάμαι θα λάβουν την ίδια απάντηση. Εγώ ήρθα εδώ για να συζητήσω μαζί σας για τα θέματα αρμοδιότητάς μου. Αν ε, επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά μου. Γιατί η χρηματοδότηση τρομοκρατιών είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα και καλωσορίζω τη δουλειά που κάνετε σε αυτό το τομέα. Θέλω το ταχύτερο δυνατόν ναι, να ε, υποβάλω ε, προτάσεις, ε, σας το λέω προς ενημέρωση, για την, προτάσεις για την ποινικοποίηση, για την κατάσχεση προσόδων από παράνομες ενέργειες, παράνομες ροές χρημάτων, για να προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε λοιπόν αυτή την χρηματοδότηση των τρομοκρατών και φυσικά αυτό ε, σχετίζεται με το θέμα των καταπιστευμάτων και επειδή θα ορκιστώ στη θέση του Επιτρόπου θα, ε, θα εκπληρώσω αυτό το ρόλο και δεν θα εκπροσωπώ την ευρωτανική κυβέρνηση. Ο κύριος Τζέριτ Πάτων από το EFTD. Εδώ είμαι. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω γιατί η Βρετανία ορίζει έναν επίτροπο καθώς ο τελευταίος έπρεπε να παρατηθεί ε, και πριν 12 εβδομάδες είχαμε ένα δημοψήφισμα ο Βρετανικός λαός αποφάσισε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ακούγοντάς σας απόψε ακούγεται σαν να γίνονται οι δουλειές όπως συνήθως ε, είπατε ότι σε αυτό το ρόλο πρέπει να δώσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν όρκο ανεξαρτησίας και φυσικά δεν θα πρέπει να εργαστεί ότι θα πρέπει να εργαστείτε για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του Ενωμένου Βασιλείου και δεν θα πρέπει να λάβετε εντολές από την Βρετανική κυβέρνηση. Μας ε, είπατε ε, ότι έχετε δει, μας έχω δύο ερωτήσει αν ε, τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης του Βασιλείου συγκρούνται ποια θα εξυπηρετήσετε και πώς πιστεύετε, πόσο πιστεύετε ότι θα διαρκέσουν τα καθήκοντά σας ε, καθώς πρόκειται οποιαδήποτε στιγμή να εγκαταλείψει ε, η Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός αν κυρία Μέη δεν εννοεί ότι θα προβεί στο Brexit και τελικά ουσιαστικά η ο δικός σας ορισμός ε, εδώ θα δείξει κάτι τέτοιο. Δεν συμφωνώ απόλυτα αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά κάποιο τρόπο τον ορισμό μου ότι έχει να κάνει με τα ευρύτερα θέματα της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Δεν ε, θα παρουσιάσω ότι θα υπερασπίσω τις θέσεις της Βρετανικής κυβέρνησης απόψε, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός Μέη ήταν απολύτως ε, σαφής για το σεβασμό των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος. Πόσο καιρό θα είμαι εδώ ως αποτέλεσμα αυτού. Αυτός είναι ένας άλλος ε, ευθύς τρόπος να μου ζητάτε να κάνω μία πρόβλεψη για τις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θα μπορέσω να κάνω κάποιο σχόλιο για την διαδικασία των διαπραγματεύσεων που δεν έχει ξεκινήσει μάλιστα επισήμως. Η ερώτηση τώρα για τον όρκο. Εγώ το παίρνω πάρα πολύ σοβαρά και θα σεβαστώ τον όρκο μου. Όπως σωστά είπατε, αυτό σημαίνει ότι θα είμαι απολύτως ανεξάρτητος στη διεξαγωγή των καθηκόντων μου και ούτε θα ζητήσω, ούτε θα δεκτώ οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε άλλο όργανο ή οντότητα. Έτσι εγώ θα συμπεριφερθώ ως μέλος του Σώματος των Επιτρόπων. Ερώτηση υπέρθουν ε, γνωστό εκ μέρους ε, της κυρίας Άτκισον από το ΙΕΝΕΦ. Καλώς ορίσατε. Κύριε Σερ Τζούλιαν, χαίρομαι που η θητεία σας θα είναι εξίσου σύντομη με τη δική μου. Ε, θα επαναλάβω τα όσα είπε ο συνάδελφος. Πραγματικά εμένα με ενοχλεί το ότι παίρνετε αυτή τη θέση μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και εσείς εργάζεστε για τους 65 εκατομμύρια Βρετανούς που κατά πλειοψηφία ψήφισαν να φύγουν από εδώ. Δεν έχετε καμία υποχρέωση σε αυτό εδώ το μέρος. Σε εμάς είστε υπόλογος, για εμάς δουλεύετε. Και χαίρομαι, χαίρομαι που συμφωνείτε πως η ασφάλεια είναι εθνική αρμοδιότητα. Αλλά αν ακούσετε κάποιες συζητήσεις εδώ μέσα, ε, τι ακούμε, ανοιχτά σύνορα, ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων. Συμφωνείτε. Συμφωνείτε ότι οι τζιχαντιστές δεν θα συμφωνήσουν, δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνείτε πως πλήτεται η εθνική ασφάλεια της Ουγγαρίας, γιατί εδώ μέσα είμαστε τόσο ανίκανοι να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Συμφωνείτε με τα όσα έκανε ο Βίκτορ Όρμπαν και θα πρέπει να επαναληφθεί Um, uh, thank you. Um, uh, if... Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ειλικρινά δεν εκπροσωπώ εγώ την Βρετανική κυβέρνηση. Δεν είναι αυτή η βάση της απόψινής μας συζήτησης. Εάν με επιβεβαιώσετε σε αυτή την θέση, θα ορκιστώ χωρίς κανένα πρόβλημα και θα τηρήσω αυτόν τον όρκο. Και τότε θα εργαστώ για το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον και για λογαριασμό όλων των Ευρωπαίων πολιτών, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβανομένων και αυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι να φύγει. Και όταν φύγει, προφανώς και εγώ δεν θα συνεχίσω να εργάζομαι εδώ πέρα. Για το θέμα της ε, ασφάλειας και το εάν εδώ μέσα αυτό το μέρος μπορεί να βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι τόσο σημαντική αυτή η δουλειά. Αυτό προσπάθησα να πω. Συμφωνώ πως οι τζιχαντιστές, ε, τρομοκράτες δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό πρέπει να πολεμήσουμε τους τζιχαντιστές τρομοκράτες και να ενισχύσουμε την άμυνά μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και στα όσα άσχημα επιθυμούν για εμάς. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Περνάμε στην ερώτηση ε, υπαριθμών 9. Και να σας ευχαριστήσω για το ότι τηρήσατε το χρονοδιάγραμμα και παρακαλώ έτσι να είστε και στη συνέχεια. Ερώτηση παριθμών 9, κύριο Σιζόφσκι. Ευχαριστούμε κύριε Κίνη για την ε, παρουσίαση. Ελπίζω τα, να μιλάω αγγλικά τόσο καλά όσο εσείς γαλλικά. Πιστεύετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εμπλακεί στη διαδικασία εναρμόνισης ε, για τα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης ε, αφού αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πιστεύετε για το opt-out και τις διαπραγματεύσεις ε, για το Brexit. Ε? Μπορεί δηλαδή να προκύψει μια νέα εταιρική σχέση για αυτά τα ζητήματα. E Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση από πλευρά του ΕΛΚ. Παρακαλώ απαντήστε κύριε Κίνγκ. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα που έχω όταν προσπαθώ να σας δώσω μια διαρθρωμένη απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι και πάλι με... μου ζητάτε να συζητήσουμε τις ε, πολιτικές και τις θέσεις της Βρετανικής κυβέρνησης και να ε, κάνω εγώ υποθέσεις για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την έκβασή της. Επιτρέψτε μου λοιπόν να περιορίσω την απάντησή μου στο εξής. Όπως είπα επανειλημμένα, πιστεύω πως αυτές οι απειλές και οι προκλήσεις στα θέματα ασφαλείας είναι κοινέ και ε, αγγίζουν όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Η Βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει και αυτό θα κάνει, θα τηρήσει την έκβαση του δημοψηφίσματος. Εξακολουθεί όμως το Λονδίνο να είναι δύο ώρες με το τρένο από τις Βρυξέλλες και από το Παρίσι. Οι τζιχαντιστές δεν κάνουν καμία διάκριση ανάμεσα στις Βρυξέλλες, το Παρίσι και το Λονδίνο. Κάνουν καμία διάκριση ανάμεσα στις σχέσεις που έχει μια χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις ίδιες σχέσεις θα έχουμε και φυσικά θα έχουμε κοινά συμφέροντα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές. Ευχαριστούμε. Δεύτερη ερώτηση από τους σοσιαλιστές. Η Μάριον Λόρστιν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ξέρετε διριστέντα επίτροπε, θα ασχοληθείτε με τα διαλειτουργικά συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ άλλων βάσει του χαρτοφυλακίου σα και στι γραπτέ σα απαντήσει είπατε θα ενθαρρύνετε την ομάδα υψηλού επίπεδου για τα συστήματα ασφαλεία. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο μπορείτε να μας πείτε ακριβώς ποια συνεργασία μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, εσείς ποιες ιδέες θα αναδείξετε σε προτεραιότητα και συγκεκριμένα. Αυτή την ομάδα εμπειρογνωμών θα την υποστηρίξετε για να δημιουργηθεί μια σούπερ βάση δεδομένων, ένα κοινό αποθετήριο ευρωπαϊκό δεδομένων, αντί για το Eurodac και άλλα συστήματα που είναι ξεχωριστές βάσεις, εθνικές βάσεις δεδομένων. Ποιο συγκεκριμένα μπορείτε να μας πείτε τι είδους κινδύνους διαβλέπετε για μια τέτοια υπέρβαση δεδομένων όταν το εξετάζουμε αυτό το θέμα από την οπτική γωνία της προστασίας των ατοπικών δεδομένων θα θέλατε, είπατε, να εξασφαλίσετε μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα ασφάλειας και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων. στην περίπτωση της υπερβάσης δεδομένων, τι πιστεύετε για αυτή την ισορροπία. Ευχαριστώ. Ε, ναι, σας ευχαριστώ για την, την ερώτηση και το πλαίσιο στο οποίο τη θέσατε. Ε, έχετε εις βάθος γνώσεις για την προστασία δεδομένων και το εκτιμώ. Το ανέφερα στις παρατηρήσεις μου διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η υψηλή ομάδα εμπρογνωμόνων και πραγματεύεται ζητήματα κέρια σημασία. Ελπίζω να κάνουν γοργά βήματα, να συνεχίσουν την εργασία τους το 2017 και αν εγώ μπορώ να κάνω κάτι για να τους ε, βοηθήσω σε αυτή τη χρονική κλίμακα θα το κάνω. Η νομική, τεχνική και επιχειρησιακή διάσταση όλων αυτών των ζητημάτων είναι αυτό που τους απασχολεί. Και επειδή δεν υπάρχει μόνο το μοντέλο στο οποίο αναφερθήκατε, υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα εναλλακτικών λύσεων, έχοντας αυτού κατά νου, ε, ελπίζω τα θεμελιώδη δικαιώματα και συγκεκριμένα η προστασία των ατομικών δομένων, ελπίζω να είναι στον πυρήνα των εργασιών τους. Υπάρχει ένας τρόπος έτσι ε, να λάβουμε υπόψη αυτά ε, τα δεδομένα, διότι το σύστημα είναι όσο τα δεδομένα που εισαγάγουμε και τα δεδομένα που βγαίνουν από αυτό το σύστημα. Οπότε θα δούμε αν ε, διακριτά συστήματα μπορούν να είναι διαλειτουργικά, μπορούν να επικοινωνούν. Και από ό,τι κατάλαβα, μία από τι εναλλακτικέ που θα εξετάσουν αυτή που αναφέρατε, αυτή τη κοινή βάση δεδομένων. Όποια εναλλακτική και αν εξετάσουν, όποια σύσταση και αν ε, ε, καταθέσουν, είμαι πεπισμένο ότι θα τηρήσουν τους κανόνες για την προστασία των ατομικών δεδομένων και με, τα χαράς να, σε συστηματική βάση να σε ενημερώνουν για την πρόοδο των εργασιών αυτής της ψηλής όμως εμπειρογνωμών. Ερώτηση 11. Χέλγα Στίβεν, δεύτερη ερώτηση του ECR. Παρακαλώ. Sir Julian King, do you believe... Πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη μέσω ε, εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρέπει να συνεργαστούν με τους παρόχους πρισιών διαδικτύου προκειμένου να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες ε, και να αποτρέψουν ε, επιθέσεις Είχαμε μια πρόσφατη γνωμοδότηση του δικαστηρίου σε σχέση με τη συμφωνία PNR Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Επίση, η Κομισιόν σκοπεύει να παρουσιάσει προτάσει για τη συλλογή δεδομένων PNR για τα πλοία και τα τρένα, καθώ και αυτά αρχίζουν να, να γίνονται στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. σε σχέση με τη συνεργασία με τους παρόχους ε, υπηρεσιών διαδικτύου. Νομίζω ότι αυτός είναι ένα σημαντικός τομέα. Έχει πολλές διαφορετικές πτυχές. Μία πτυχή που λαμβάνω ιδιαίτερα υπόψη στο πλαίσιο της καταπολέμησης της οικοποίησης, της ρητορικής του μίσους και της ανεπιθύμητης προπαγάνδας των τρομοκρατών είναι το όλο δίκτυο δίκτυο του τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο, τι είναι εκούσιο, τι είναι υποχρεωτικό και πώς μπορούμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό διάλογο με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου για τα θέματα αυτά. Και σας ευχαριστώ που ε, κληρονομώ ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για το διαδίκτυο όπου συμμετέχουν ε, τα κράτη-μέλη και εμπειρογνώμονε του διαδικτύου για να συζητούν κάποια από αυτά τα θέματα. Θέλω να δω αν μπορούμε να αναπτύξουμε την εργασία μας και να την προωθήσουμε. Ρωτήσατε και για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης Καναδά για τα PNR και την γνωμοδότηση του δικαστηρίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την ε, έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο, αλλά προκύψουν θέματα. Θα πρέπει να εργαστούμε στα πλαίσια της απόφασης σε ό,τι αφορά τώρα την επέκταση του PNR, το δεδομένο του καταλόγων επιβατών. Όταν συζητήθηκε το θέμα αυτό, αποφασίστηκε σε εκείνο το στάδιο να μην συμπεριληφθούν ή να μην επεκτείνουμε τα δεδομένα PNR για να καλύψουμε και άλλα είδη μεταφορών όπως σιδηροδρομικές, χερσαίες μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές και αυτό ε, φαντάζομαι ήταν εν μέρη επειδή αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερα δεδομένα. Και κάποιες φορές ε, αυτή η πάροχοι ούτως ή άλλως δεν ε, συνέλεγαν αυτά τα δεδομένα κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Τώρα, αν ξαναδούμε την εφαρμογή του PNR και φυσικά υπάρχει ένα πρόγραμμα προς αναθεώρηση, αφού θα τεθεί σε σχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να έχουμε κάποια διδάγματα από το πώς τέθηκε σε εφαρμογή και να δούμε αν μπορεί να επεκταθεί. Αλλά οποιαδήποτε επέκταση θα πρέπει ε, να γίνει σύμφωνα με την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα, σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια. Ευχαριστώ. Έχουμε καθυστερήσει κατά 9 λεπτά, έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έχετε κατά νου το χρόνο που περνάει. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση είναι από την κυρία Γκρίσμπερκ, πάλι από τους φιλελευθέρους. Ε, κύριε, ε, τα επίτροπε, μεταξύ των ε, στρατηγικών καθηκόντων που προτείνονται για αυτό το χαρτοφυλάκιο αναφέρεται και το θέμα της κυβερνοασφάλειας και της ενισχυμένης ψηφιακής ασφάλειας. Πολύ ε, λίγο έχουν ε, αναπτυχθεί όμως αυτά τα θέματα αυτά. Όπως ξέρετε, οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο και πριν ε, λίγες μέρες ε, στη χώρα μου, στη Γαλλία, ε, αντιμετωπίστηκε, λύθηκε μια επίθεση εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες. Ήθελα να μου πείτε πώς θα δράσετε σε αυτό το με δεύτερον. Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών online είναι πραγματική μάστεγα παρά την οδηγία του 2011 και η οδηγία αυτή μας δείχνει τα ωριά της καθημερινά αν ε, η ε, αν εσείς οριστείτε ως Επίτροπος, πώς θα δράσετε, τι δράση θα αναλάβετε σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να εκφράσω την ε, πάση αλληλεγγύη μου στη Γαλλία αυτή την περίοδο γιατί πράγματι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά με τις επιθέσεις που πολύ συχνά ανακύπτουν. Σε ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και θέλω ως προτεραιότητα να θέσω την εφαρμογή των οδηγία που αφορά τα συστήματα πληροφορικής θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν σχέδια για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, να κάνουν κάποιες έρευνες για να αντιμετωπίζουν ε, κάποια περιστατικά και χαιρετίζω το γεγονός ότι υπάρχει τώρα συμφωνία για ε, μια νέα σχέση, εταιρική σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα μεταξύ δηλαδή των επιχειρήσεων και των δημοσίων αρχών για να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω εργασία σε αυτό το τομέα. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει αυτό το έργο για τα παιδιά και για την εφαρμογή της οδηγίας του 2011. Εγώ ε, γνωρίζω πόσο σημαντική είναι αυτή η οδηγία, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο φάκελος. Θα ήθελα ως Επιτροπή να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας και θα πρέπει σύντομα να παρουσιάσουμε μια αναφορά. Ζητώ συγγνώμη που έχουμε καθυστερήσει κάπω, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνει εντό του έτου. Έχουμε τώρα την δεύτερη ερώτηση από την κυρία Σπινέλη. Παρθμό 13. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ βρίσκομαι. Στις 23 Αυγούστου, οι Υπουργοί Εσωτερικών Γαλλίας και Γερμανίας ανακοίνωσαν ότι στη Σύνοδο της Βρατισλάβα θα ζητήσουν από την Κομισιόν δηλαδή και σε, από εσά, κύριε Κίνγκ, μία οδηγία για τον encryption, για την κρυπτογράφηση που θα υποχρέουν εταιρείε όπως η WhatsApp ή η Telegram να μειώσουν τα πρότυπα της κρυπτογράφησης ή να βάλουν κάποιες πίσω πόρτες ε, προκειμένου η αστυνομία να μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Η πρόταση δέχτηκε κριτική από τους υποστηρικτές της ε, προστασίας ιδιωτικής ζωής και από την Γαλλική Αρχή Προστασίας των Δεδομένων. Δηλαδή, ε, αυτή η αφαίρεση της κρυπτογράφησης ε, θέτει σε κινδύνους τους πολίτες σε άλλες μορφές τρομοκρατίας, ε, πολύ πιο απελητικές από την τρομοκρατία των κρομοκρατών. Ποιες εγγυήσεις εσείς θα δώσετε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των πολιτών και δεύτερον, δεν πιστεύετε ότι ο τρομοκράτης θα υπερβεί τα εμπόδια χρησιμοποιώντας ή και δημιουργώντας κάποιες εναλλακτικές ε, τέτοιες εφαρμογές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που θέτετε αυτό το σημαντικό θέμα. είναι κρίσιμο το διαδίκτυο σε όλες τις πτυχές της ζωής μας και στην ιδιωτική μας ζωή, όπως φαίνεται από όλες τις τελευταίες ερωτήσεις και φυσικά έχουμε ιδιωτική ζωή και online και offline. Και η ασφαλής επικοινωνία και η κρυπτογράφηση είναι τμήμα αυτού του κόσμου και είναι τμήμα της ιδιωτικής ζωής που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Επίσης, Ισχύει ότι κάποιοι πολύ κακοί άνθρωποι χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, οι τρομοκράτες και πράγματι η επίθεση που μόλις αναφέρθηκε που πρόσφατα αποκαλύφθηκε και στη Γαλλία χρησιμοποίησε και πάλι μια γνωστή συσκευή κρυπτογράφησης για το σχεδιασμό. Όμως δεν είναι μόνο οι τρομοκράτες, ε, αλλά και εγκληματίες που χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση. Επομένως δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Δεν είμαι πεπισμένος ε, ότι ουσιαστικά υπάρχει το μαγικό ραβδί που θα δώσει τη λύση. Ε, εγώ ε, ουσιαστικά δεν θεωρώ ότι αν βάλουμε ουσιαστικά κάποιες πίσω πόρτες πρόσβασης κάτι τέτοιο θα μας κάνει πιο ασφαλείς. Θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί και εναντίον μας. Και από τρίτα μέρη δεν είναι λοιπόν απλό το ζήτημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων, το Internet Forum που συμμετέχουν και τα κρατημέλη αλλά και εμπειρογνώμονε που θα διερευνήσουν αυτό το ζήτημα. Εγώ θα ήθελα να το πράξω αυτό και θα ήθελα να του ζητήσω να μας ε, παρουσιάσουν κάποιε συστάσεις που ευχαριστώ θα συζητήσω μαζί σα. 14 second Greens question from για τον ε, κύριο Λάμπερτ, 14η ερώτηση. Ευχαριστώ, θα ήθελα να σχολιάσω τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Αναφερθήκατε στον Καναδά, αλλά φυσικά η Τουρκία, το Αφγανιστάν, μια σειρά από χώρες. Και αν κοιτάξουμε τώρα αυτό το θέμα της συνεργασίας και της ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αποτελεσματικότητας, το βλέπουμε και σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις έκτακτες επιδόσεις ε, και την εμπλοκή κάποιων κρατών μελών. Εκεί τέθησαν πάρα πολλά ερωτηματικά για την ε, λογοδοσία και την ε, αποτελεσματικότητα της παράκαμψης διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές αρχές συνεργασίας με τρίτες χώρες και πώς θα εξασφαλίσετε μια αυξημένη διαφάνεια για το σεβασμό αυτών των αρχών. Απάντηση. Ε, οι αρχές που για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι ταυτόσιμες με τις αρχές που θέλω να διέπουν τη συνεργασία με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το λόγο δράσεις που εκπίπτουν διεθνούς δικαίου και καταφανώς παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα όπως ε, οι ε, εκδόσεις πρέπει άνευ επιφυλάξεων να κατακριθούν όπως έχει γίνει και επανειλημμένα. Η αποτελεσματικότητα όμως δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει να βρούμε μια κοινή προσέγγιση για την ε, τήρηση του διεθνούς δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία μας με τρίτες χώρες. Για στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίας όπως ε, αυτή με τις είπα, αν αυτό έχετε στο μυαλό σας, Μπορώ να πω ότι εν μέρη χάρη σε προσπάθειες ευρωβουλευτών και ειδικότερα μελών της Επιτροπής Νομίζω ότι είναι πιο ισότιμη η σχέση σε σχέση με το παρελθόν. Τέλεια δεν είναι, δεν μπορώ να το ισχυριστώ, όμως ε, είναι θετική η κατεύθυνση που ακολουθούμε. Και αν θέλετε, η, η προστασία, ε, η αποκατάσταση και η συμφωνία, ε, η Γενική Συμφωνία, αυτό το τρίπτυχο μας επιτρέπει να τηρήσουμε τις αρχές που θέλουμε να ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που περιμένουν να ισχύσουν και για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Λόρα Φεράρα από το EFTD. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Κίνγκ. Θα είστε υπεύθυνο για την εσωτερική ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, η επιστολή του κυρίου Γιούνκερ ε, αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τους υπόλοιπους επιτρόπους και στις όμως δεν καταλαβαίνω που ακριβώς είναι τα όρια της δικής σας εντολής και που αρχίζει ε, η αρμοδιότητα των συναδέλφων σας και αναφέρομαι κυρίως στην κυρία Γιούροβα και στον κύριο Ευρωμόπουλο και στις δηλώσεις σας ε, πέρα από κάποιες αναφορές στην τρομοκρατία δεν βρήκα συγκεκριμένες αναφορές συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που είναι ένα φαινόμενο επίσης πολύ σημαντικό και είναι σε, τόσο σημαντικό όσο και η τρομοκρατία. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω, σκοπεύει η Κομισιόν να αντιμετωπίσει το θέμα της ασφάλειας χωρίς να αντιμετωπίσει στο σύνολό του το οργανωμένο έγκλημα γιατί το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το 2013 θετήθηκε μια ανακοίνωση από την Κομισιόν και πρόκειται να, από, συγγνώμη, ένα ψήφισμα από το Κοινοβούλιο και θα υιοθετήσει κι άλλο σε σχέση με τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν θα υπάρχουν κάποιες συστάσεις και ποια θα είναι η σειρά προτεραιοτήτων που θα θέσετε. Ευχαριστώ. Ε, ε, thank ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ έστω και σύντομα για... στο θέμα του οργανωμένου κλίματος που ξέρω πως σας απασχολεί σε αυτή την Επιτροπή. Η έκθεσή σας θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να έχουμε μια συζήτηση εις βάθος για αυτό το θέμα και πραγματικά την αναμένω με ανυπομονησία κάποιες από τις προτεραιότητες ε, που χαράξατε εσείς με τους ε, συναδέλφους, δηλαδή η αντιμετώπιση της διαφθοράς, το θέμα της ε, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και οι νέες καινοτόμες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, το περιβαλλοντικό έγκλημα, η διακίνηση μορφών άγνεων ζώων. Αξίζει πραγματικά να το δούμε πιο στενά. Και καθώς περνάμε σε μια επανεξέταση του κύκλου πολιτικής, εγώ θα ήθελα να βασιστούμε στην επιτυχία του προηγούμενου, της προηγούμενης περίοδου, από το 2013 μέχρι σήμερα, να δούμε ζητήματα όπως η πλαστογραφία, την κυβερνοασφάλεια και τα όπλα και να τα ανανεώσουμε για να λάβουμε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις. Οπωσδήποτε θα ήθελα να χρησιμοποιήσω όλα τα υφιστάμενα μέσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στις υπηρεσίες για να δούμε αυτό το ζήτημα και να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, για να γίνει αυτό βασικό στοιχείο του διαλόγου με τρίτες χώρες για το πώς ελπίζω να εργαστώ όπως σας είπα αυτό θα πρέπει να το δούμε στην ε, πράξη. Σκοπεύω να αποτελέσω μέλος μιας ομάδας και να συνεργαστώ στενά με τους επιτρόπους σε αυτά τα ζητήματα και θα είμαι υπόλογος σε εσάς για την διάσταση της ασφάλειας. Η ερώτηση 16 είναι η δεύτερη ερώτηση του ΙΕΝΕΦ από την κυρία Τκίνσον. Και πάλι, για να δούμε τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπατε πως ε, το, τα σύνορα του Ηνωμένου ε, έχουμε πλέον ε, και του Ηνωμένου Βασιλείου στο Γκάρντινορ και τους έχω συναντήσει και μου έχουν πει τους φόβους τους γιατί εάν συνέβαινε μια ασφάλεια μια, με συγχωρείτε, επίθεση τζιχαντιστική υπήρχε κίνδυνος και είχαν μάλιστα έρθει σε επαφή με την Υπουργό Εσωτερικών τότε Τερέζα Μέη να περάσει ο έλεγχο των διαβατηρίων μέσα στην ασφαλή περιοχή, γιατί θεωρούσαν ότι κινδύνευαν οι ίδιοι. Ε, σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να προστατεύσουμε τους ε, Βρετανούς συνοριοφύλακες. Όπως σας λέω, απερίφραστα, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ε, όχι, συμφωνώ οπωσδήποτε. Η προστασία των Βρετανών πολιτών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς στο επίκεντρο της δουλειά ε, Δεν αποφεύγω την ερώτηση, αλλά και πάλι σας λέω δεν εκπροσωπώ τη Βρετανική κυβέρνηση εδώ απόψε. Οπωσδήποτε θα αντλήσω από τις εμπειρίες μου αυτές ε, στον νέο μου ρόλο και μία τέτοια εμπειρία είναι η πολύ στενή συνεργασία που είχα επί σειρά ετών και εντατικά τους τελευταίους μήνες με την Βρετανική Συνοριοφυλακή κάνουν εξαιρετική δουλειά και αν και ξεφεύγει λίγο από το σημερινό μας θέμα θα ήθελα να χαιρετήσω την δουλειά που κάνουν στη Βόρεια Γαλλία και βοηθούν τους ε, ταξιδιώτες να μετακινούνται μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και της Υπηρετικής Ευρώπης. Εάν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να στηρίξουμε την αποτελεσματική δράση στα σύνορα, οπωσδήποτε θα ξεκινήσω αμέσως σε συνεργασία με τον κύριο Αβραμόπουλο. Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση από το ΕΛΚΑ από την κυρία Βόζενμπεργκ. Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Κίνγκ. Έχετε δηλώσει ότι μέσα στις προ... προτεραιότητές σας είναι ο αποκλεισμός πρόσβασης τρομοκρατών στη χρηματοδότηση. Αυτό το επαναλάβατε και σήμερα, αναφερόμενο σε κάποιες επικείμενες πρωτοβουλίες από την Επιτροπή. Με αυτό το δεδομένο, παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν, είναι, αν προτίθεστε να φέρετε νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που θα καλύπτει παραδείγματος χάρη πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής ανάλογου αντίστοιχου προγράμματος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Νομίζω πώς αυτό σχετίζεται και με την προηγούμενη ερώτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας. Οι διευθετήσεις με τη ΣΥΠΑ που αναφέρατε και πάλι βεβαίως εδράζονται στην ε, Europol και είναι πολύ αποτελεσματικές. Ακόμα και αν κάποιος μετακινεί μεγάλα ποσά, καμιά φορά το να ιχνηλατήσουμε την κίνηση αυτών των κεφαλαίων είναι πολύ χρήσιμο για τις έρευνες. Υπήρχαν κυριολεκτικά εκατοντάδες ίχνη από αυτό το σύστημα μετά τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες και το Παρίσι και ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Τώρα, ρωτήσατε εάν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμπληρωθεί από μια διευθέτηση ανάλογη μεταξύ των κρατών μελών ε, στο πλαίσιο της ε, ΣΕΠΑ, της περιοχής πληρωμών. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι την τελευταία φορά που εξετάστηκε αυτό, αυτή η ιδέα, πριν από λίγα χρόνια, δεν δόθηκε συνέχεια από την Κομισιόν, αλλά κατά την άποψή μου η απειλή πλέον έχει αλλάξει, όπως είπα και συζητάμε σε όλη αυτή την ακρόαση. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε ξανά την κατάσταση και να καταλήξουμε σε κάποιες επιλογές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτή τη στιγμή, για να τις συζητήσουμε εντός του έτους. Thank you. Question Σας ευχαριστώ. Ερώτηση 18. Πίτερ Ντερμούλερη, τρίτη ερώτηση των σοσιαλιστών. Εντάξει. Ναι, έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, σύμφωνα με την επιστολή για την ανάθεση κάθε κόντων που σα έστειλε ο κ. Γιούνκερ. Θα είστε υπεύθυνο για την αναβάθμιση του κέντρου αντιδρομοκρατίας της Europol. Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτό. Δεύτερον, μετά τι αποκαλύψει Snowden και τα ευρωπαϊκά αιτήματα για την απαγόρευση και την μείωση της κρυπτογράφησης, τι άποψη έχετε γι' αυτό. Και τρίτον, πρόσφατα Είχαμε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά κάποιων μέτρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παραδείγματος χάρη η Συμφωνία Ασφαλούς Λιμένα. Πώς θα διασφαλίσετε εσείς στο χαρτοφυλάκιό σας ότι η Κομισιόν δεν θα υιοθετήσει νομοθεσία η οποία αργότερα θα ανατραπεί από το Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω πρώτα απ' όλα την δεύτερη ερώτηση, γιατί αν κατάλαβα καλά, Δεν έχω και πολλά να προσθέσω στα όσα είπα για την κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι βασικό κομμάτι του διαδικτύου. Εξυπηρετεί πολύ καλούς σκοπούς όσον αφορά την ιδιωτική ζωή. Επίσης όμως γίνεται κατάχρηση της από τρομοκράτες ε, και παιδόφιλους. Δεν υπάρχει κάποια εύκολη απάντηση ή απλή λύση για να το σταματήσουμε αυτό και θέλω να υπάρξει ένας διάλογος με τους παρόχους ε, του διαδικτύου και άλλους για να έχουμε κάποιες ιδέες προς συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πλησιάσουμε καν σε συστάσεις. Ε, τώρα, για το κέντρο της αντιδρομοκρατίας και την ενίσχυση της Europol, νομίζω πως έχουμε μια ευκαιρία τώρα, την οποία πρέπει πραγματικά να αρπάξουμε από τα μαλλιά. Και θα συνεργαστώ με τον Διευθυντή της Europol για να είμαστε σίγουροι ότι θα έχει τους απαραίτητους πόρους, χρηματοδότηση και εμπειρογνωμοσύνη για να γίνει το αντιτρομοκρατικό κέντρο στο δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να αποσπάσουν εκεί ειδικού, να μοιραστούν την εμπειρία τους και βέβαια θα θέλαμε να βασιστούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελεσματικής συνεργασίας όπως παραδείγματος χάρη την ε, επιχείρηση που έλαβε χώρα μετά την επίθεση στο Παρίσι για να έχουμε μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου. Τώρα, για το πώς θα συντάξουμε καλύτερη νομοθεσία, ελπίζω να με βοηθήσετε εσείς σε αυτό, όπου αυτό απαιτείται, γιατί όπως είπα πρέπει να εφαρμόσουμε και κάποια πράγματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Αλλά εάν απαιτούνται νέα μέτρα, οπωσδήποτε ε, δεν θα διστάσουμε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πραγματικά ποιοτική νομοθεσία η οποία θα μπορεί να αντέξει στο χρόνο και βεβαίως, όπως είπα, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σχετικές δομές. Πολύ λεπτομερής ε, αυτή η ερώτηση. Θα σας παρακαλούσα πάντως, συνάδελφοι, να προσπαθήσετε να σεβαστείτε τα χρονικά όρια. Περνάμε στην τρίτη ερώτηση του ECR από την κυρία Χαλάχο. Από τον κύριο Χαλάχο. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας ε, για δύο νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια. Καταρχήν η οδηγία για τα πυροβόλα όπλα σύμφωνα με τον Επίτροπο θέλει να κόψει την πρόσβαση των τρομοκρατών στα πυροβολά Στην πραγματικότητα όμως η πρόταση ε, επιτίθεται ουσιαστικά στην νομίμη οπλοκατοχή και ε, με ουσιαστικά μία σύνδεση με την ε, παράνομη οπλοκατοχή. Εσείς πιστεύετε ότι σέβεται αυτή η πρόταση την αναλογικότητα, την αναγκαιότητα ε, της αρχές αυτές και δεύτερον έχουμε και το θέμα του συστήματος εισόδου-εξόδου το Κοινοβούλιο ανησυχεί για την πρόσβαση των διοκτικών αρχών στα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται. Οι εθνικές αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτή η πρόσβαση έχει προστιθέμενη αξία, αλλά κάποιοι στο Κοινοβούλιο δεν είναι πεπισμένοι. Πώς βλέπετε την ισορροπία μεταξύ της ανταλλαγής πληροφοριών για ε, στόχους ε, επιβολής του νόμου και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ευχαριστώ. Κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις ε, φαίνονται να έρχονται από πολλές πλευρές. Ε, κάποιοι συνάδελφοι ρωτούν δύο-τρεις ερωτήσεις ε, και ουσιαστικά τις θέτεται αυτές σε 20-30 δευτερόλεπτα, αλλά αν ο πρέπει να απαντήσει χρειάζεται περισσότερο χρήμα, τέλος πάντων. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Κίνκ. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικέ οι ερωτήσεις. Βέβαια, ξέρετε τελικά ποιο είναι το σκορ, θα συνεχίσουμε έτσι. Έτσι θα είναι η κατάσταση όταν <laughs> παρουσιάσετε οποίο μας, θα ξέρετε κύριε Κίνγκ. Λοιπόν, για τα πυροβολά όπλα. Accordingly, sorry, everyone. Συγγνώμη αν επιβεβαιωθείτε, αν όλα πάνε καλά και φυσικά σας εγκρίνουν οι συντονιστές. Σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση για τα πυροβολά όπλα. Νομίζω ότι το είπα στην ανακτήρια δήλωσή μου. Για μένα η πρώτη πρόκληση είναι η παράνομη ε, εμπορία όπλων, το λαθρεμπόριο όπλων. Και θα ήθελα η Ευρωπόλ, το σύστημα της Interpol, το σύστημα της Ευρωπόλ να συνεργαστεί με τους εταίρους από τις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι γίνεται ήδη καλή δουλειά στο διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί και ίσως και να επεκταθεί σε άλλες χώρες για να καταπολεμήσουμε το παράνομο λαθρεμπόριο όπλων. Αν καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο των όπλων, ε, νομίζω ότι θα ουσιαστικά θα έχουμε και κάποιε αυστηρότερε διευθετήσεις για την όμιμη απλοκατοχή. Και καλωσορίζω το γεγονό ότι ω ε, μέρος αυτού έχουν ληφθεί ήδη αποφάσει για την ε, επανέναρξη, δηλαδή για να δούμε και πάλι το θέμα των όπλων που έχουν απενεργοποιηθεί. Κάποιες φορές αυτά τα όπλα που έχουν απενεργοποιηθεί επανενεργοποιούνται και χρησιμοποιούνται. Όμως θα πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι και στις ε, ανησυχίες που ακούγονται από την νόμιμη χρήση όπλων από τους πολίτες μας. Ε, θα ήθελα να το δούμε αυτό το ζήτημα και να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Τώρα για τα ΕΦΗ e e σύνορα και για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Είναι μια νέα πρόταση, ε, αντικατατρίζει εκτεταμένη συζήτηση. Εγώ θα συνεργαστώ πολύ στενά με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο Καθώ είναι ο αρμόδιο και θα την προωθήσει. Και σας είπα, χωρί να μπερδεύουμε τα πράγματα, υπάρχει και μια διάσταση ασφαλεία σε ό,τι αφορά του ελέγχου που κάνουμε στα σύνορά μας. Και όσο το κάνουμε αυτό συνεκτικά με το πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του σεβασμού των αρχών της αναγκαιότητας, αναλογικότητας κτλ. Νομίζω ότι θα δράσουμε στο στα πλαίσιο. Λοιπόν, ε, έχουμε την ερώτηση, τρίτη ερώτηση για τους φιλελευθέρους, τον κύριο Λουί Μισελ. Κύριε Οριστέντα Επίτροπε, μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που είναι διαπραγμάτευση σε τριμερή διάλογο, Νομίζω ότι έχουμε μια σοβαρή ευκαιρία να καλύψουμε τα κενά του νέου συστήματος του Ευρωπαϊκού PNR. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά αυτόματη ανταλλαγή των δεδομένων PNR των υπόπτων ή των ε, ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί δυνάμει με την οδηγία για την καταπλήρωση τρομοκρατίας. Αυτό θα μας επιτρέψει πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Θα υποστηρίξετε αυτή την πρόταση εσείς. Επίσης, η ανταλλαγή δεδομένων έχει κάποια όρια. Ε, πώς, παραδείγματο χάρη, εσείς θα δράσετε έτσι ώστε τα δεδομένα PNR να αναλύονται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θα ήταν σκόπιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε μια κοινή ανάλυση κινδύνου αυτών των δεδομένων, αναρμονίζοντα τον ορισμό της ύποπτης συμπεριφοράς, παραδείγματο χάρη. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρετε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, Πριν να θέσουμε την ερώτηση για την κοινή ανάλυση αυτού του συστήματος. Θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ο πρώτος στόχος που θα είχα θα ήταν να συνεργαστώ στενά με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να συστήσουν ε, τις PIU αυτές τις μονάδες γιατί δεν τίθεται καν το ζήτημα χωρίς αυτές. Και από όσο γνωρίζω, τώρα έχουμε δύο ή τρία κρατημέλη που είναι σε θέση να ζητήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας ακόμη. Αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και το ελπίζω φυσικά σε αυτό το σημείο, βεβαίως θα υπάρχει το εξή ερώτημα. Πώς θα συνεργαστούμε ε, αποτελεσματικά. Πώς θα συνεργαστούν αποτελεσματικά οι σε αυτό το κρατών μελών. Και ευχαρίστω ε, θα καταρτίζαμε βέλτιστε πρακτικές, κατευθυντήρε γραμμές για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, σε όλα αυτά τα ζητήματα βρίσκω ότι δρώντας το πλαίσιο των συνθηκών θα πρέπει να βάλουμε τη δυνατά μας ε, για να έχουμε ουσιαστικά κοινό επιμερισμό των ευθυνών. Τώρα, για το τι μπορούμε να κάνουμε κατά της τρομοκρατίας. Ελπίζω ότι τώρα θα μπορέσουμε να κινηθούμε γρήγορα όλοι μαζί. Γιατί πρέπει να δούμε όλες τις στοιχείες, το θέμα του ταξιδιού ή το θέμα της εκπαίδευσης, των τρομοκρατών ε, ή το θέμα τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατία. όλα αυτά θα πρέπει να συμπιώσουμε πρόοδο. Σα ευχαριστώ. 21η ερώτηση από την ΚΟΕ, από την κυρία Άντερσον. Σας ευχαριστώ. Πώς ε, έχετε αναλύσει, πώς έχετε σκεφτεί το θέμα της Ιρλανδίας μετά από το Brexit ουσιαστικά λένε σήμερα ότι δεν θα υπάρχει σκλήρινση ε, σε ό,τι αφορά το θέμα των συνόρων. Εσείς πώς θα εργαστείτε για να αποτρέψετε πιθανές εγκληματικές δραστηριότητες σε ένα εξωτερικό σύνορο μελλοντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα ε, διασφαλίσετε αυτή την πίσω πότρα πριν να φύγετε. Φυσικά ε, θα προετοιμάσετε όλα αυτά τα θέματα πριν να φύγετε, όμως πώς θα διασφαλίσετε την Τελωνιακή Ένωση και ουσιαστικά ε, να μην ε, υπάρχουν ουσιαστικά κάποια μειονεκτήματα, να μπαίνουν ε, κάποια από την Βρετανία μέσα σε ένα κράτο μέλο και να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα διασφαλίσετε ότι όλη αυτή η προστασία, η διασυνοριακή, ουσιαστικά δεν θα οδηγήσει σε διχοτόμηση της Ιρλανδίας, κάτι που θα ήταν απόλυτη καταστροφή. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει μόνο με τη θέση της κυβέρνησης να πει υπηρετώ αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως σε λίγο δεν θα την υπηρετώ και θα προσπαθήσω να αντιβατήσω γιατί θίγει κάποιες ευθύνες, κάποια καθήκοντα που θα έχω στον νέο μου ρόλο. Εγώ ξέρω προσωπικά πόσο σημαντική είναι η ζωή ε, για όλους τους ανθρώπους ε, που κατοικούν βορείως και νοτίως αυτού του συνόρου. Εγώ το έχω περάσει, έχω περάσει αυτά τα σύνορα, έχω φίλους που ζουν και από τις δύο πλευρές και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Δουβλίνο, στο Μπέλφαστ και στο Λονδίνο να γίνει μια προσπάθεια να βρούμε έναν τρόπο να αποφύγουμε όλα αυτά τα μειονεκτήματα που αναφέρατε. Όμως αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και των 27 κρατών μελών. Και επιλέγω να μην το σχολιάσω αυτό σήμερα και ελπίζω να καταλάβετε γιατί. Είναι κάτι για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην ερώτηση 22 από τους Πρασίνους. Είναι η τρίτη ερώτηση. Είναι Φίλιπ Άρμπλεχτ. Σας ευχαριστώ. Ήδη ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες νομίζω απαντήθηκαν επαρκώς. Θα ήθελα εγώ να προσθέσω την πτυχή τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη. Όπως ε, ήδη ε, παρουσιάσατε την θέση σας εντός της Κομισιόν και το πώς θα εργαστείτε εντός της Κομισιόν και με το Κοινοβούλιο. Αλλά πώς θα μπορέσουμε να έχουμε εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων στα κράτη-μέλη και πώς ε, θα έχετε την στήριξη των κρατών μελών για ένα κοινό σχέδιο δράσης όταν μιλάμε για την Ένωση Ασφαλείας και ειδικά όσον αφορά μέτρα καταπολέμησης της ρίσοσπαστικοποίησης όπου εμείς θεωρούμε πως πρέπει να τεθεί το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές στα κρατη Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχουν δύο μέρη σε αυτή την ερώτηση. Το πρώτο είναι πώς θα οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη με τις εθνικές αρχές και το άλλο είναι τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε σε διάφορα πλαίσια, συχνά με τις εθνικές αρχές, συχνά χωρίς αυτές, με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και άλλους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στην εκπαίδευση, στις φυλακές όπως είπατε και αλλού που αντιμετωπίζουν τη ζωσπαστικοποίηση. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε με τα κράτη-μέλη, όπως είπα στην αρχή, υπάρχει ένας ξεκάθαρος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συνθήκων για να ενθαρρύνουμε, να βοηθήσουμε, να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα και να επιβάλλουμε αν αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης υπάρχει ένας ρόλος για να ορίσουμε προδιαγραφές και να παραμερίσουμε εμπόδια στην συνεργασία. Αναφέρθηκα ήδη ακριβώς στην ε, ερευνητική αυτή ε, ομάδα η οποία έχει στόχο να ε, αφαιρέσει εμπόδια από την, στην συνεργασία. Επίσης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη ακριβώς με συγχωρείτε τα θεσμικά όργανα να βοηθήσουν ε, εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα με τα κράτη-μέλη και να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, όπως είπα, μεταξύ των κρατών μελών, αλλά όχι μόνο εκεί. Και αυτό θα ήθελα να τονίσω στην απάντησή μου. Πιστεύω πως ε, η πιο επιτυχής ε, δράση κατά της ριζοσπαστικοποίηση δεν γίνεται από τα κράτη, αλλά από την κοινωνία των πολιτών και γι' αυτό πρέπει να τους χρηματοδοτήσουμε, να δώσουμε την απαραίτητη προγνωμοσύνη και να έχουν επαφές σε ολόκληρη την Ευρώπη έτσι ώστε να έρθουν αυτοί σε επαφή και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε μια ερώτηση από την Επιτροπή Άφετ, ο κύριος Πάσκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζουμε όλοι πως υπάρχει μια τάση να ενσωματώνουμε τις εσωτερικές με τις εξωτερικές πτυχές της ασφαλείας. Και αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό της ε, κατάστασης ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε. Και συγκεκριμένα τώρα εσείς θα βρεθείτε σε μία θέση ακριβώς στην καρδιά αυτής της, ε, του συνδυασμού θα έλεγα των δύο πτυχών έχετε σκεφτεί καθόλου συγκεκριμένα την συνεργασία αυτή αφενός ε, με ε, επιτρόπους ε, με την είπατε εκπρόσωπο, με επιτρόπους που ασχολούνται με τα εξωτερικά και με τον συντονισμό του, του Κέντρου. Ναι, ευχαριστώ. Έχω ξεκινήσει τις συναντήσεις μας και ακριβώς το το ζήτημα το οποίο θέσατε. Δηλαδή υπάρχουν δύο πτυχές εδώ. Η εσωτερική και η εξωτερική ε, ασφάλεια και σε πολλούς τομείς πρέπει να ενισχύσουμε και τις δύο πτυχές. Και η μία ενισχύει την άλλη αν το πετύχουμε σωστά. Οπότε εγώ θα θέλω να συνεργαστώ με την Αντιπρόεδρο την κυρία Μογκερίνη και τους συναδέλφους της Κομισιόν όσο το δυνατόν πιο στενά, έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ανησυχίες της ασφάλειας, εσωτερικής, εξωτερικής και κοινή ασφάλειας, στον διάλογο με τις τρίτες χώρες. Παραδείγματο χάρη, σκέφτομαι τη συνεργασία που μπορούμε να έχουμε σε ζητήματα αντιμετώπισης ε, του βίαιου εξτρεμισμού, το τι μπορούν να κάνουν για να μας βοηθήσουν στις προσπάθειες ε, από ριζοσπαστικοποίησης. Προφανώς το προφανές η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ακριβώ η ανάγκη καταπολέμησης του λαθρεμπορίου όπλων. Αυτοί είναι κάποιοι τομεί στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε και υπάρχουν κάποιες ε, διαρθρωτικές σχέσεις πολύ σημαντικές. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι μια βελτιωμένη δομή της σχέσης μας με τη ΣΥΠΑ και θεωρώ πως και γενικώ και σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα ο συνάδελφος που καθόταν στην θέση σας ρώτησε για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η συνεργασία μας με τρίτες χώρες έχει μεγάλη σημασία για την εσωτερική μας ασφάλεια. Ευχαριστώ. 23. Τρίτη ερώτηση από, τον, ε, από το EFTD, ο κύριος Μπάτν. Ευχαριστώ, Κλοντ Τζούλεν ήρθατε ή θα είσαστε εδώ πέρα για να βοηθήσετε στη σύσταση μια Ένωση για την Ασφαλεία. Για το 2013 είπε η Europol, πολιτικέ για το ελεύθερο εμπόριο και οι μετακίνησει ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντικείμενο εκμετάλλευση για την οργανωμένη εγκληματικότητα. Στο, στα εσωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν υπάρχει ελευθερία μετακίνηση, έχουμε μικρότερε πιθανότητε ανείχνευση. Ε, συμφωνείτε ότι έχουν δημιουργηθεί έτσι μιμίζωνα προβλήματα ασφάλειας για την Ένωση και για τα κράτη-μέλη. Η προτινόμενη Ένωση για την Ασφάλεια δεν είναι άλλο ένα παράδειγμα που δημιουργεί ως προβλήμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρότασης λύσης ε, που όμως συνεπάγεται με αυξημένες αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κινητήριος δίνουμε πίσω από την Ένωση για την Ασφάλεια μήπως είναι η ανάγκη να διατηρήσουμε το, οικοδόμημα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ζωντανό παρά για να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ειλικρινά πιστεύω ότι η κινητήριο δύναμη και σίγουρα τα κίνητρα τα δικά μου, εάν επιβεβαιωθώ σε αυτή τη θέση, είναι να κρατήσουμε ασφαλείς τους πολίτες μας. Η κινητήριο δύναμη είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της κυβερνο... κυβερνοεγκληματικότητας, της κυβερνοτρομοκρατίας. Ελπίζω να προέκυψε με σαφήνεια αυτό από τις απαντήσεις που σας έδωσα. Σε αυτό αποβλέπω και αυτός είναι ο στόχος ε, των καθηκόντων μου. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα οποιασδήποτε συνεργασίας με εσάς, με τα κράτη-μέλη ή με την κοινωνία των πολιτών για να φτιάξουμε την ε, Ένωση για την Ασφάλεια. Και πάλι, οι χειρότερες ε, περιπτώσεις ε, που αντιμετωπίζουμε, οι χείριστες τρομοκρατικές ε, προθέσεις, ουσιαστικά δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας σύνορα Σέγγεν ή μη Σέγγεν. Επιτίθενται κατά ενός τρόπου ζωής και από αυτό πρέπει να προστατευτούμε. Ερώτηση 25, τέταρτη ερώτηση από το έλικο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ. Κύριε Κίνγκ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω με πάσα ειλικρίνεια και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Η Ένωση ασφάλεια. είναι μια ωραία φράση που θα τη βιώσουμε για κάποιο καιρό. Το βέβαιο όμως είναι αυτό που λέει το άρθρο 4. Εσείς το παραθέσετε. Η αρμοδιότητα είναι των κρατών μελών. Εδώ όμως είμαστε στα πλαίσια της συνεργασίας. Η Ευρωπόλ βάσει ε, του κανονισμού του 2017 θα είναι ένα μέσο συνεργασίας ε, για τα κρατημέλη. Και θα σας δώσω και μία είδηση. Δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν σχετικά οι συνεργάτες σας. Η ανακοίνωση της Κομισιόν της 20 Απριλίου θεσπίζει για την εφαρμογή του θεματολογίου για την ασφάλεια ότι τον Οκτώβριο του 2016, το, φθι, το, το φθινόπωρο μάλλον του 2016, μέσα σε 90 μέρες πρέπει να παρουσιάσετε πρωτοβουλίες για να ενισχύσετε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της Ευρωπόλη. Και θα πρέπει να παρουσιάσετε συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό επιμένω στις ερωτήσεις, αλλά με ένα συγκεκριμένο τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά το δικό σας κριτήριο, ποια μακροπρόθεσμα και πρόθεσμα πέτρα θα μας παρουσιάσετε με 90 μέρες για να ενισχύσετε το κέντρο και πώς θα βελτιώσετε την ε, ικανότητα σχεδιασμού και πρόληψης και τέλος η σχέση μεταξύ του ECTC και του Τμήματος ε, Ανάλυσης Στρατηγικών Πληροφοριών της κυρίας Μογκερίνη. Δεν μιλάω για δήλωση αρχών, αλλά πώς θα γίνει ο συντονισμός. Αυτό με ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη. Uh, thank you. Um... Ευχαριστώ και ελπίζω να μπορέσω και εγώ να επωφεληθώ από την πραγματογνωμοσύνη και την εμπειρία σας για να εργαστούμε μελλοντικά σε αυτό το τομέα και να προωθήσουμε τα αισθήματα που μας ενδιαφέρουν. Ε, χαιρόμαστε Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση που μου κάνατε. Σίγουρα θα ε, καταθέσουμε νέες ιδέες, θα κάνουμε προτάσεις και επίσης σίγουρα είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το νέο νομικό πλαίσιο που αρχίζει να ισχύει το Μάιο του 2017 και πρέπει να προετοιμαστούμε ήδη από τώρα γι' αυτό. να είμαστε θέση λοιπόν, στο μέτρο που μπορώ, αναφίβολα θα υποστηρίξω ένθερμα τη θα υποστηρίξω το πλαίσιο της πολιτικής, θα υποστηρίξω μέσω χρηματοδότησης προσωπικού, είτε πρόκειται για νέο προσωπικό, ε, νέους πόρους ε, για τη Europol, καλύτερη απόσπαση εθνικών πραγματογνωμών προς την Europol και επί τη βάση που έχω δει χρειάζεται αναβάθμιση με 80-90 υπαλλήλους για να επιτελεστούν τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Europol και θέλω να ε, προσφέρω συγκεκριμένα σε αυτή την προσπάθεια. γιατί η λειτουργική δυναμικότητα, φυσικά αυτό είναι στο πίνον της εργασίας του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, ε, διότι μιλάμε για το ίντερνετ, τη δράση στο διαδίκτυο, για τη χρηματοδότηση για το συνεχιζόμενο διάλογο με τις εθνικές αρχές. Θέλω να ενισχύσω λοιπόν τις καλές εμπειρίες που είχαμε για την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών και να ενισχύσουμε αυτό το ρόλο. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι πολλά τα, αυτά που πρέπει να κάνει ε, για το λαθρεμπόριο και για το κυβερνοέγκλημα η Europol, οπότε μην ξεχνάμε το θέμα της επιχειρησιακής ε, δυναμικότητας της Europol και ξαναλέω θα την υποστηρίξω και όπως είπα και σε προηγούμενη απάντηση, ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω, τόσο ώστε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες περισσότερο, που προκύπτουν φυσικά από το Europol και το Eurojust. Α, και το τελευταίο που είπατε, Ε, ναι, ανάμεσα στο Ένσεν και το ACTC είναι οι δύο όψεις ε, του ιδίου νομίσματος, ε, διότι μιλάμε για εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Ε, συνάδελφοι, πρέπει να επανέλθουμε στο, στα μονόλεπτα και δίλεπτα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους ακόμη. Ερώτημα 26 τέταρτο. Ε, ερώτημα από τους σοσιαλιστές Τάνια Φαγιών. Ευχαριστώ συνάδελφοι, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τις νέες τεχνολογίες για την ασφάλεια. Βάσει του ρόλου σας, πώς θα εξασφαλίζετε ότι θα χρηματοδοτηθεί έρευνα ε, σε αυτό το τομέα, διότι δεν χρειαζόμαστε μόνο ειδικού, όπως αναφέρετε και εσείς στις απαντήσεις σας, ε, αλλά ε, είναι η λιδία λήθος και για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, για την ανταλλαγή συγκεκριμένα βιομετρικών δεδομένων. Τι πιστεύετε, ε, για την ανείχνευση, αναγνώριση προσώπων και σχετικές άλλες τεχνολογίες για την ασφάλεια. Πόσα θα αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις τέτοιων προγραμμάτων και νέων τεχνολογικών μέσων επί της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Απάντηση. Νομίζω ότι η χρηματοδότηση για την έρευνα και η σχέση της με τους στόχους που έχουμε θέσει στον τομέα της ασφάλειας έχει αυξανόμενη σημασία. Εγώ σε μεγάλο βαθμό υποστήριξα ε, κάποια ρηξικέλευθα βήματα που έχουν γίνει στο μέτρο της έρευνας για τα θέματα ασφάλειας. Φερρυπίν, υπάρχει ένα κομμάτι που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της έρευνας, όπου οι πρόδρομοι απενεργοποιούνται οι πρόδρομες ουσίες, δηλαδή δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ε, πρόδρομες ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές δημοκρατικές επιθέσεις. Επίσης κάτι άλλο που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την βελτίωση του, της λειτουργίας του ραντάρ σε συνεργασία με την επιχείρηση Σοφία. Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στον τομέα της ασφάλειας και τα ερευνητικά προγράμματα και θέλω να ενθαρρύνω αυτήν την αμφίδρομη σχέση. Όπως είπατε σωστά, για να ενθαρρύνουμε την ενερεύνα, κατά νου θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το πλαίσιο που, στο οποίο αναφερθήκαμε πολλά και σήμερα, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ε, βασικό σε θεμέλιος λήθος ε, του έργου μας στην Ένωση. Με τους συναδέλφους επιτρόπους μου με, που άμεσα ε, έχουν άμεση αρμοδιότητα για την ε, επόμενη, τα επόμενα ερευνητικά προγράμματα. Αυτό τον στόχο θα υλοποιήσω. Ε, ECR, τέταρτη ερώτηση, Μόνικα μακβει Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω. Έχουμε δύο φακέλους για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενίσχυση των ελεγχών για τις βάσει δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρόκειται για τροποποίηση του κώδικα Σέγγιν ε, ουσιαστικά. Έχουμε διάσταση απόψεων γι' αυτό και ρωτώ ποιο είναι ο ρόλος σας ε, διότι κατεπήγοντα χρειαζόμαστε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους πολίτες μας, χρειαζόμαστε καλύτερη διαχείριση και θωράκιση των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκής Ένωση, Πιστεύετε ότι συστηματική έλεγχη και αποτελεσματική χρήση όλων των ε, σημαντικών βάσεων δεδομένων θα αυξήσει, θα ενισχύσει την ασφάλεια θα καταστήσει αποτελεσματικότερα τα σύνορά μας ε, για την ε, για να αμυνθούμε κατά ιονή τρομοκρατών. Δεύτερη ερώτηση. Πώς βελτιώνατε την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών και τις αρχές επιβολής νόμου στα κράτη-μέλη και συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και πυριών στους αρμόδιους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπαρκτό πρόβλημα αυτό. κακή συνεργασία, λειψή συνεργασία, γολένουσα συνεργασία. Πάντηση. Ευχαριστώ. Για την ασφαλεία στα εξωτερικά μας σύνορα. Όπως σας είπα νωρίτερα, πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορες στρώματα ασφάλειας που χρειαζόμαστε και σίγουρα ένα από αυτά που πρέπει να ενισχύσουμε είναι τα εξωτερικά μας σύνορα. Θέλω να συνεργαστώ στενά με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και άλλους από το Σώμα Επιτρόπων για τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις, στις οποίες και αναφερθήκατε, κύριε Μακοβέ. Πιστεύω πως ε, συντρέχει λόγος να περάσουμε στη φάση των συστηματικών ελέγχων. Νομίζω ότι αιτιολογείται, όπως είπα και νωρίτερα, η εξέταση εναλλακτικών ελέγχων που μπορούν να γίνουν στα εξωτερικά σύνορα, κυρίως για επικός χωρών και όντως συμφωνώ πως πρέπει να μας απασχολήσει πώς αποτελεσματικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που απορρέουν ε, περιορίζοντας τους στόχους χρήσης και έτσι προστατεύοντας τα ατομικά δικαιώματα. Με του όπως σας είπα, πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα και να καταθέσουμε συγκεκριμένες συστάσεις. Για το θέμα της ε, συνεργασίας ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής νόμου, συμφωνώ μαζί σας ότι είναι δύσκολη η συνεργασία ορισμένε φορές και εσωτερικό ενός κράτους μέλους, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι ήταν αριστή η συνεργασία ανάμεσα στη Europol και τις ε, γαλλικές και βελγικές αρχές για την επιχείρηση που κατέληξε σε συγκεκριμένη πρόοδο και δόθη συνέχεια ε, με αποτελεσματικό τρόπο στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Ε, οικοδομώντα επί αυτή τη συνεργασία των βελτίστων πρακτικών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προσκόμματα που ενδεχομένω ε, ενίοτε ανακύπτουν στη συνεργασία αυτών των αρχών. Ε, Μόρα, συνάδελφοι, δεν ξέρω, έχουμε, επειδή είναι Δευτέρα, έχουμε αργήσει, μήπω εγώ φταίω, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, Σοφία Ιντβέλτ, ερώτηση 28. Κυρία Ιντβέλτ, καλώ ορίσατε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την έμφαση που δίνετε στην παραγωγή αποτελεσμάτων και την υπόσχεσή σας να αξιολογήσετε την τρομοκρατική στρατηγική. Θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι οι στρατηγικές μας μέχρι τώρα ήταν επιτυχημένες ή αποτυχημένες. Είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας τα τελευταία 50 χρόνια ή όχι και πιστεύετε ότι υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να καταργηθούν. Μιλάμε για νέα μέτρα. Βλέπετε κάποια που θα μπορούσαν να καταργηθούν. Δεύτερη ερώτηση. Φαίνεται να προτείνεται ότι η κριτική των ΗΠΑ μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνεργασία μας. Νομίζω ότι είναι κάπως περίεργο αυτό, γιατί εντός ε, των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο έντονη η κριτική που ασκείται. Παραδείγματο χάρη, αναφέρομαι στην ουσία Στέν και στην Επιτροπή τη. Τι θα κάνετε εσεί για να πετύχετε λογοδοσία για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο με τη CIA. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αξιολόγηση. Αυτό το οποίο θεωρώ είναι ο τρόπος στον οποίο μάθαμε να αντιδρούμε σε κάποιες από αυτές τις απειλές ε, και επιθέσεις έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν είναι ο ίδιος με αυτό το οποίο συνέβη πριν από 15 χρόνια αμέσως μετά τις επιθέσεις και προσωπικά είναι κάτι το θετικό για, θεωρώ εγώ γιατί θεωρώ πως είναι πιο έξυπνη η αντιμετώπιση πώς το αξιολογώ όμως πώς θα ήταν τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα αν δεν είχαμε κάνει τα όσα κάναμε. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ δύσκολα αλλά θεωρώ πως εάν ε, πρέπει να κάνουμε μια καλή αξιολόγηση, θα πρέπει στο πλαίσιο του της καλύτερης νομοθεσίας που διατρέχει το έργο αυτής της Κομισιόν και με το οποίο συμφωνώ θα πρέπει να έχουμε βεβαίως και μια αίσθηση αναλογικότητας και για τα όσα θα κάνουμε από εδώ και μπρος αλλά και όταν επανεξετάζουμε τα όσα κάναμε στο παρελθόν σε άλλους τομείς αρμοδιότητας κομισιών κάποια πράγματα έχουν ανακληθεί και καταργηθεί και δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει να εφαρμοστεί και εδώ κάτι τέτοιο. Για την κριτική στις είπα Ναι, μάλλον όχι. Λάθος. Ήταν αυτό το οποίο είπα. Ε, θεωρώ πως ε, κάποια από την κριτική η οποία ασκήθηκε και από αυτή την Επιτροπή και από αυτό το Κοινοβουλίο βοήθησε σημαντικά να βελτιωθεί η κατάσταση στη ΣΥΠΑ και η σχέση μας με τη ΣΥΠΑ γιατί μετά από πράγματα τα οποία εσείς και άλλοι σε αυτήν την Επιτροπή θέσατε πιστικά καταφέραμε να έχουμε την δομή που έχουμε με αυστηρότερους κανόνες για πρόσβαση στα δεδομένα, έναν μεσολαβητή, μια δυνατότητα προσφυγής, δεν υπάρχουν μαζικές, στοχευμένες και χονδρικές ε, παροχές στοιχείων κτλ. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να είμαστε πολύ ε, αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ. Ερώτηση 29, τέταρτη ερώτηση της Γκουε, η Μαρή Κριστίν Βερζιά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Καλησπέρα σας, κύριε Κίνγκ. Ευχαριστούμε και για την εξαιρετική γνώση των γαλλικών. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της βάσης δεδομένων και στη διαλειτουργικότητα των βάσεων αυτών. Από τότε που εργάζομαι επί του θέματος αυτού, θεωρώ ότι το κύριο πρόβλημα είναι η υλοποίηση από τα κράτη-μέλη και δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όσο εσείς για τη συνεργασία μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας, αν και κάπως έχει βελτιωθεί. Και πάλι πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες και αν ήταν καλύτερη, ίσως είχαμε αποφύγει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα μακριά από την επιμερισμένη ευθύνη την οποία επιθυμείτε. Τα κράτη-μέλη ουσιαστικά παραμένουν στις δικές τους αρμοδιότητες ε, ουσιαστικά τα θέματα ασφαλείας δεν είναι μόνο ε, διεθνή αλλά είναι και διεθνή εντός, υπερεθνικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι βάζουμε ε, όλο και πιο μακριά το πύχη και όλο πιο ψηλά αλλά εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δεν τεταφή σύνορα και το σύστημα εισόδου-εξόδου, ε, ουσιαστικά το είχαμε σχεδιάσει για τις τουριστικές ροές και τώρα μιλάμε για έλεγχο των συνόρων και το οργανωμένο έγκλημα και τα δύο μπορούμε να τα επενέσουμε, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε τι κάνουμε και νομίζω ότι επιγόντως χρειαζόμαστε πραγματική αξιολόγηση του συνόλου αυτών των βάσεων δεδομένων με τους συγκεκριμένους στόχους. Τελειώνω, Πρόεδρε με τους συγκεκριμένους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή, πώς εξελίχθηκαν, γιατί και ποια είναι τα αποτελέσματα σε τεχνικό και νομικό επίπεδο, κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να μπορούμε να αξιολογούμε τις δράσεις μας και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουμε θέσει σε εφαρμογή. Και είμαι έτοιμος μαζί σας να συνεργαστώ για κάτι τέτοιο. Επίσης συμφωνώ ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και πρέπει να είναι ένα θέμα προτεραιότητας θα πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερα τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Παραδείγματο χάρη, έχω κατά νου και συγγνώμη αν κάνω λάθο με τα αρχικά, αλλά έχω κατά νου την συνθήκη του ΠΡΟΥΜ, όπου έχουμε τρεις πτυχές και συμμετέχουν 18-20 κράτη-μέλη τα οποία πράγματι μπορούν να θέσουν ε, σε εφαρμογή τις συμφωνίες αυτές. Και οι τρεις πτυχές, για αυτές τις τρεις πτυχές υπάρχουν όμως κρατημέλη που δεν μπορούν να το πράξουν αυτό. Επίσης, έχω κατά νου αυτό, δεν σχετίζεται με το σύστημα πληροφορικής, <clears throat> αλλά έχω κατά νου και το θέμα των πρόδρομων ουσιών για τα κρυκτικά. όπου δεν εφαρμόζονται οι κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιδιώξουμε τους στόχους που όλοι έχουμε θέσει από κοινού. Σας ευχαριστώ. Είμαστε 20 λεπτά πίσω στο χρόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, για Κοιτάξτε τώρα, αν θέλει ο καθένας να μιλάει 30 δευτερόλεπτα παραπάνω, εγώ δεν συμφωνώ. Όταν κάποιος ξεπερνά το χρόνο θα χτυπά το σφυράκι. Και αυτό αφορά και τον οριστέντα επίτροπο. Δίνετε όλοι στα δύο λεπτά. Περνάμε στον κύριο Τερικάμπρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κίνγκ, Μία αποστολή σας θα είναι, μία αποστολή της ε, εσωτερικής σας μονάδας θα είναι η ταυτοποίηση τρομοκρατικού ε, περιεχομένου. Πώς όμως θα εγγυηθείτε ότι θα ταυτοποιηθεί μόνο τρομοκρατικό περιεχόμενο και μόνο τέτοιο θα σβήνεται. Και σημαντικότερο, ποιο, πότε και πώς θα καθορίσει σαφώς το τι εστί τρομοκρατικό περιεχόμενο. Πώς θα διασφαλίσετε ότι η Europol ή η μονάδα αυτή θα συμμορφώνεται με την αρχή του περιορισμού του στόχου όταν αναλαμβάνει τέτοια καθήκοντα. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ αφενός ε, ε, κηρυγματών των μίσους και παρότρινση σε βίες πράξεις που είναι παράνομο και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του νόμου και κάποιον πραγματικά θα έλεγα αποκουστικού τρομοκρατικού περιεχομένου η προπαγάνδα σε οποία όμως δεν είναι προπαγάνδα μίσους αλλά είναι πολύ δυσάρεστη και αυτή ακριβώς η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε και πρέπει να μας απασχολήσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι τώρα έχουμε κάποιες δομές που εξετάζουν το ζήτημα με πλήρη διαφάνεια και κοιτάνε την συνεργασία με παρόχους διαδικτύου που από τη δική τους την πλευρά συνεργάζονται με διαφάνεια και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό. Δεν έχω κάποια έτοιμη απάντηση στην ερώτησή σας γιατί δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το εφαρμόσουμε αυτό. Αλλά όταν βλέπουμε πράγματα τα οποία πραγματικά είναι επιλήψιμα, σε κάποιες περιπτώσεις θα κατεβαίνουν και σε άλλες περιπτώσεις, και είμαι ανοιχτό εδώ πέρα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε να υπάρχουν εναλλακτικά μηνύματα και αφηγήσει και αφηγήματα, τα οποία θα είναι επίσης διαθέσιμα. Είναι και τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να δούμε με τους παρόχους του διαδικτύου, αλλά νομίζω πως ε, το οφείλουμε στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης της ρίζοσπαστικοποίησης να δώσουμε στον κόσμο επιλογή, διαφορετικά μηνύματα και να τους ενθαρρύνουμε να εξασκήσουν ακριβώς ε, την λογική τους. Σας ευχαριστώ. Ερώτηση 31 Beatrice von Storch, Sir Julian. Η αποστολή σας θα είναι οπωσδήποτε η Ένωση της Ασφαλείας και σύμφωνα με τον Γιούνκερ εδώ πέρα θα πρέπει να εφαρμόσετε την ε, σχετική ατζέντα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν την ελευθερία, ακούσαμε την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα, τα δεδομένα αεροπορικών επιβατών. Οπότε θα αφαιρέσετε κάποιε ελευθερίε και λέτε ότι σε αντάλλαγμα θα του προσφέρετε ασφάλεια. Ε, έχει ξαναδοκιμαστεί αυτό και δεν λειτουργήσε. Είστε λοιπόν αρμόδιος για αυτό, αλλά στην εντολή σας, στην επιστολή αυτή, δεν εμφανίζεται ούτε μία φορά η λέξη σύνορα, μόνο η λέξη διασυνοριακά εγκλήματα μέτρα όπως ε, η ευθυροποίηση της ε, οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα είναι κατανοητά. Πόσο σημαντική είναι για σας η προστασία των συνόρων. Uh, uh, um, and I, uh, Ευχαριστώ και συμφωνώ όπως ε, είπαμε ότι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε είναι κάποιες από αυτές τις απειλές ε, είναι στα σύνορα. Γιατί ε, από τη φύση τους, όπως σωστά λέτε, μιλάμε για διασυνοριακές απειλές. Και ε, βεβαίως αν τα αντιμετωπίσουμε στα σύνορα θα τις διαταράξουμε καλύτερα αυτές τις δραστηριότητες. Γι' αυτό ελπίζω ότι απάντησα σε αρκετές ερωτήσεις, σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον, για το πώς θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους. Θα λάβουμε υπόψη τα μέτρα τα οποία υπάρχουν ήδη ή σχεδιάζουμε να τεθούν ενισχύ σύντομα την διάσταση της ασφάλειας στα σύνορα. Και εδώ πέρα θα είμαι υπόλογος σε εσάς για την αποτελεσματικότητά τους ε, και την ε, συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες γιατί όπως ε, και εσείς έτσι και εγώ δεν θέλω να αφαιρούμε ελευθερίες. Σας ευχαριστώ. Η πέμπτη ερώτηση του ΕΛΚ, η συντονιστής, η κυρία Χολμάιερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε επίτροπε, κύριε Κίνγκ, σε αντίθεση με τον ε, κύριο Φανστόρκ δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι συνοριακοί φράχτες, αλλά ο καλύτερος συντονισμός των αστυνομιών διασυνοριακά. Έχουμε ένα τελείως ανομοιογενές ε, πεδίο εδώ πέρα, δηλαδή άλλοι έχουν τελείως διαφορετικούς χρόνους αντίδρασης ε, και πεδία και περιοχές ευθύνης ε, και πώς ακριβώς θα προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα για την διασφάλιση διασυνοριακά της ασφάλειας των πολιτών μέσω της συνεργασίας των αστυνομιών. Thank you very much. Um, I entirely agree and a number of questions. Σας ευχαριστώ και σε διάφορες απαντήσεις σας είπα ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές ε, πρέπει ε, ανάντι να δράσετε ε, ορισμένε φορές ε, στα σύνορα ή και στο εσωτερικό των συνόρων μέσα στα πλαίσια μια κοινή προσπάθεια Και έχουμε συζητήσει ήδη για τους διαφόρους τρόπους με τους μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Για την ενθάρρυνση τη διασυνοριακή συνεργασίας, σημαντικό τμήμα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα μέσα και τα συστήματά μας, αλλά και οι φορείς να μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά μαζί, ούτω ώστε με αποτελεσματικότητα να βοηθούν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιώντας την νομοθεσία ή άλλα κίνητρα που υπάρχουν για την άρση των προσκομμάτων ε, για τη συνεργασία. Πρότυπο, παραδείγματος χάρη, αν υπάρξει αμοιβή αναγνώριση των προτύπων ε, λειτουργίας, αυτό μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία. Είπα νωρίτερα ότι υπάρχει η εντολή έρευνας ε, που έπεται. Πολύ καλό παράδειγμα αποτελεσματικής δράσης για να έχουμε μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων στα κράτη-μέλη, διευκολύνοντας ταχεία δράση σε περίπτωση δίωξης. Μπορούμε λοιπόν με διάφορους τρόπους να σημειώσουμε πρόοδο. Ερώτηση 34, πέμπτη από τη σοσιαλιστές Τάνια Φαγιών. Ευχαριστούμε κύριε Κίνγκ. Είναι ε, η επίκαιρη ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών έχει κέρια σημασία για την αποτελεσματική συνεργασία των αρχών επιβολής νόμους, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως είδαμε συγκεκριμένα στην πράξη πώς τα κράτη-μέλη ε, δεν χρησιμοποιούν ε, μέσα που υπάρχουν, όπως το ΣΥΣ ή η απόφαση πριν, αποτελεσματικά. Το 2005 προσάρμοσε το Συμβούλιο μια απόφαση όπου είναι λεπτομερείς οι διατάξεις για την υποχρέωση κρατών μάλλον για την ανταλλαγή πληροφοριών για τρομοκρατικές επιθέσεις, ανταλλαγή τόσο με κράτη-μέλη όσο και με οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτηση. Ποια βήματα θα κάνετε συγκεκριμένα ούτως ώστε έγκαιρα να γίνεται αποτελεσματικά η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί και η ποιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται. Θα κινήσετε διαδικασία επί παραβάση κατά των κρατών μελών που συστηματικά δεν πληρούν αυτή τη νομική τους υποχρέωση να ανταλλάξουν πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ε. απόφαση πριν, για το συζητήσαμε ήδη, έχουμε διάφορες ε, πιλωτικούς διαρθρωμένους διαλόγους, μια ίστατη προσπάθεια, αν θέλετε, για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν λάβει ήδη δέσμευση. Μίλησα για τις πρόδρομους ε, για τα εκρηκτικά, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Έχουμε ήδη κινήσει διαδικασία σε παραβάση. Προφανώς, αν δράσει κάποιος ε, ε ανάντι είναι πιο αποτελεσματικό και το PNR, τα στοιχεία επιβατών. Αναφερθήκαμε σε αυτό από πλευράς νομικού πλαισίου, πολύ σημαντικό. Όμως, υπάρχει πολύ πρακτική πλευρά. Τα PIUs, χωρίς τα PIUs δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα. Δύο κρατμέλη έχουν συγκεκριμένα ε, σχέδια για τις μονάδες αυτές. Μπορούμε να τα ενθαρρύνουμε με σονομικής και τεχνικής αρρωγής, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και 15 εκατομμύρια και 70 για τα επόμενα χρόνια. Οπότε δεν πρόκειται μόνο για διαδικασίες παραβάση, αλλά ναι, εκεί που χρειάζεται, ναι, γιατί όχι. 35-5 ερώτηση ECR ε, Βέστησον. Θα μιλήσω δανέζικα. Kommissærkandidat, jeg øh, Εσείς ε, θέσατε δύο συγκεκριμένα θέματα σήμερα και ουσιαστικά οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και το ΕΛΚ ε, έχουν εκφράσει την ανησυχία να γίνει η Europol ε, κάτι σαν ευρωπαϊκό FBI. Μπορείτε να μας πείτε ότι εσείς συμμερίζεστε αυτή τη φιλοδοξία. Έτσι θα πρέπει να ερμηνεύσουμε τις προσπάθειες της Κομισιόν. Επίσης, σε σχέση με το opt-out που έχει η Δανία, δεν υπάρχει συμμετοχή στη Europol, στη Eurojust, ε, στην πρόταση PNR, αν και η Δανία ανήκει στην Συμφωνία Σέγγεν. Σε αυτούς ε, τους τομείς δεν υπάρχει συμμετοχή. Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν ωφέλη, αν συμμετέχει η Δανία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τι μπορείτε να κάνετε για να διευκολύνετε αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δύο διαφορετικές ερωτήσεις και η απάντησή μου θα εξαρτηθεί από αυτά που είπαμε πολλά και σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή ότι Πολλά μπορούμε να κάνουμε, αλλά εντό του πλαισίου των συνθηκών. Και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Αυτό έλεγα μέχρι τώρα. Επομένως, η Ευρωπόλ μπορεί να υποστηρίξει αναλυτική και επιχειρησιακή δουλειά και μπορεί να προωθήσει τη συνεργασία, αλλά δεν μπορεί να είναι FBI γιατί αυτό λέγεται ξεκάθαρα στο άρθρο 88 της συνθήκης. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας για τη Δανία και για τη σχέση με την ε, Europol, με την Ευρωπόλ. Υποστηρίζω την Ευρωπόλ και ελπίζω να το αποσαφήνεις αυτό και υποστηρίζω και την ε, δέσμευση των κρατών μελών στην Ευρωπόλ, όμως εντός του πλαισίου των συνθήκων. Και όπως ξέρετε, καλύτερα από μένα, η Δανία έχει το πρωτόκολλο 22 και αυτό ρυθμίζει τη σχέση της στον τομέα. Υπήρξε δημοψήφισμα για το θέμα αυτό και επομένως πρέπει να σεβαστούμε και αυτό το δημοψήφισμα αλλά και άλλα δημοψηφίσματα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην ερώτηση 36 για την κυρία Χωσμενόφα από τις Φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τον Ιούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μία έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Ως ε, πολίτης της Βουλγαρίας χαίρομαι που θα εφαρμοστεί και στα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγιν. Στη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση η Βουλγαρία έχει ένα πολύ δύσκολο καθήκον να διαχειριστεί τα εξωτερικά στρατηγικά σύνορα της Ένωσης. Ε, και μας δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο ΣΥΣ, παραδείγματος χάρη. Επομένως, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ποια εργαλεία θα πρέπει να αναπτυχθούν για να υποστηρίξετε τις προσπάθειες της καταπολέμησης της τρομοκρατίας χωρών που έχουν εξωτερικά σύνορα αλλά δεν ανήκουν στις έγκεν Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τις προσπάθειες που καταβάλει η Βουλγαρία και την συνεισφορά της στη Europol με τη Frontex για την εκπαίδευση της ΕΠΟΛ αλλά και σε άλλους τομείς. Εγώ πραγματικά κατανοώ και βλέπω με συμπάθεια την ερώτησή σας. Η Βουλγαρία είναι στο ΣΥΣ για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, αλλά δεν συμμετέχει για άλλα θέματα μετανάστευσης. Εν τέλει, φυσικά έχει να κάνει η ερώτηση με τη συμμετοχή στη Σέγγεν και όπως ξέρετε αυτό το θέμα αφορά τα κράτη-μέλη της Σέγγεν. Όμως νομίζω ότι αυτή η ερώτηση πρέπει να τίθεται. Ξυπηρετεί πράγματι το συλλογικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά να μην συμπεριλάβουμε χώρες όπως η Βουλγαρία που βρίσκονται και στα εξωτερικά σύνορα, να μην τις συμπεριλαμβάνουμε στο σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών. Λοιπόν, έκτη ερώτηση για το ΕΛΚΟ, Κύριο Μπόνη. Κύριε υποψήφιο Πέτροπη, καθώς ε, συνεχίζεται η ψηφιακή επανάσταση και αλλάζει τον κόσμο, το έγκλημα στον κυβερνό χώρο επίσης ε, μεγενθύνεται ταχύτητα. Ε, παγκόσμια οικονομική αξία όλου του είδους του κυβερνοκλήματος ε, είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα όλα τα εγκλήματα έχουν ψηφιακές μορφές από τα χρήματα, την παράνομη εξαίρεση χρημάτων μέχρι την κακοποίηση παιδιάων οι Ευρωπαίοι ε, θα πρέπει να ενδυναμώσουν τη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα εγκλήματα με τον ίδιο τρόπο και στον κυβερνοχώρο αλλά και στην πραγματική ζωή. Έτσι λοιπόν ποιες θα είναι οι πράξεις προτεραιότητας για να καταπολεμηθεί το έγκλημα στον κυβερνοχώρο υπό αυτή την ευρία έννοια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω την ευκαιρία να επικεντρωθώ σε αυτή την πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που θα ήθελα να επιδιώξω και να δώσω έμφαση στους Αδελφου μου την Κομισιόν για το ε, έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Το ένα είναι να καταπολεμήσουμε το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το άλλο είναι να έχουμε ανθεκτικότητα ε, στον κυβερνοχώρο και όπως σας είπα θέλω να θέσω ως προτεραιότητα την εφαρμογή του, ε, της οδηγίας ε, που αφορά το δίκτυο συστημάτων πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τώρα του εγκλήματος, του επιθετικού τμήματος αυτού του θεματολογίου, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε να δυνατόν μπορούμε καλύτερα το κέντρο της Ευρωπόλ για το κυβερνό έγκλημα. Πρέπει να το ενισχύσουμε με προσωπικό και με χρηματοδότηση έτσι ώστε να μπορεί να συνεργαστεί με τις αρχές των κρατών μελών για να αντιμετωπίζει τις κυβερνοεπιθέσεις, απάτες πληρωμών και την ε, επιγραμμική σεξουαλική κακοποίηση, εκμετάλλευση όπως αναφέρεται. Και επίσης πρέπει να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα Όπως ε, είπα νωρίτερα, μόλις δημιουργήθηκε μια εταιρική σχέση ιδιωτικού δημοσίου τομέα και θα διοχετευτούν 1,8 δις στην έρευνα και στην ανάπτυξη για την καταπολέμηση του κλίματος στον κυβερνοχώρο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος και θέλω να συνεργαστώ με τους συμμετέχοντες για να αναπτυχθεί αυτό και να συνεργαστώ και με τις τρίτες χώρες για αυτά τα θέματα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα των αποδείξεων και νομίζω ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε και τη στρατηγική του 2013. Έχουμε δηλαδή πλήρη ατζέντα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Σας ευχαριστώ. Έκτη ερώτηση από τους σοσιαλιστές, ε, την Καταρίνα Κινίτσι. Ναι. Ευχαριστώ τις ε, τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις ε, ε, δεν μπορούσαν να προβλεφθούν λόγω του τρόπου που έγιναν εσείς θα αναφερθείτε και στην πρόληψη. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε κατά του βίου εξτρομισμού, όχι μόνο για την πρόληψη της ζωσπαστικοποίησης αλλά για να υπάρχουν και προγράμματα επανένταξής του στην κοινωνία. Πώς ε, αξιολογείται την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση, για την γίνεται ένα φόρουμ ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και Τέλος, για να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της επιστροφής των ξένων μαχητών, ε, θα υπάρξει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συνεργασία για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Um, thank, you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ μαζί σας πως η αντιμετώπιση της ε, ριζοσπαστικοποίησης δεν είναι μόνο θέμα προληπτικής δράσης. Είναι και δράση μετά από την ριζοσπαστικοποίηση για να αναστραφεί αυτή. Και εγώ θα ήθελα να συνεργαστώ με τα εφιστάμενα προγράμματα και δίκτυα για να καλύψουμε και τις δύο πτυχές και στην αναστροφή της ριζοσπαστικοποίησης είναι σημαντικό νομίζω να συνεργαστούμε με αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, στις ε, φύλακες όπου αντιμετωπίζουν το φαινόμενο όπως ξέρουμε τραγικά από τα γεγονότα στη Γαλλία αυτό μπορεί να είναι σοβαρή πρόκληση υπάρχουν όμως πολλές σύμβουλες ε, ειδικών ε, από ανθρώπους ε, και με στις φυλακές και με όσους εργάζονται πάνω στο αντικείμενο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντλήσουμε τα διδάγματα για συγκεκριμένη δράση κατά των ξένων μαχητών. Ελπίζω, όπως σας είπα, να διατρέχει ως νήμα τα όσα είπα απόψε το ότι η δράση θα είναι και και στα σύνορα και πίσω από τα σύνορα για να σταματήσουμε τους ε, ξένους μαχητές και άλλους ε, που προσπαθούν να μας βλάψουν. Ε, ότι θα είναι πρώτη προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. Είμαστε στην τελική ευθεία λοιπόν. Ερώτηση υπαρθμό 39, έβδομη ερώτηση του Έλκου Κέσβος. Εδώ, εδώ είμαι. Ναι, ναι, εδώ στα γερμανικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία είπατε και εντάξει κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται αλλά θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τον ψηφιακό αυτόν τον τομέα που περιλαμβάνει το κυβερνό έγκλημα αλλά και το ερώτημα πώς τελικά θα έχουμε καλύτερη χρήση τραπεζών δεδομένων με διαλειτουργικότητα. Έχω την εντύπωση πως ε, όσον αφορά την διατλαντική σχέση δεν έχουμε την καλύτερη συμπεριφορά για την συνεργασία αλλά και ότι η συνεργασία στην καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας ε, και της κυβερνο... των κυβερνοεπιθέσεων είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω Πώς θεωρείτε εσείς ότι θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτήν την σχέση, γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει κάπως διαταραχθεί, γιατί έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις ε, για θεμελιώδη δικαιώματα ή για δικαιώματα των καταναλωτών, τα οποία δεν ερμηνεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε, με ποιον τρόπο θα υπάρξει, όπως είπαμε, αυτή η συνεργασία με τις ΥΠΑ ε, και πώς θα την βελτιώσετε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τα του οίκου μας. Συμφωνώ πως υπάρχουν κάποιες στρατηγικές σχέσεις και συνεργασίες που είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του κυβερνού εγκλήματο. και όπω εξήγησα νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι όροι που διατρέχουν αυτές τις σχέσεις αλλά σε αυτόν τον τομέα νομίζω πως υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει ε, εδώ για να καταφέρουμε εμεί να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τα συστήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς την πολυπλοκότητα των κατακαιρματισμών και τα κένα αποτελεσματικά. Ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω δεν έχει αναφερθεί και μου ετέθη είναι το πώς ε, η βάση δεδομένων της Europol για την τρομοκρατία και η βάση του συστήματος δεδομένων Schengen ε, μπορούν να έχουν μια επαφή αλλά μόνο κατά περίπτωση και θα μπορούσε εδώ πέρα να υπάρχει κάποιο πρακτικό όφελο στη μεγαλύτερη διασύνδεση αυτών των δύο συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων όπου ε, έχουμε δύο βάσεις δεδομένων με πολύ παρόμοιο στόχο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα νομίζω που θα μπορούσε να κοιτάξει η ομάδα ειδικών υψηλού επίπεδου. Αλλά νομίζω πως ήμουν σαφές για το πλαίσιο και τους όρους που θα περικύκλωναν και θα, συγχωρείτε, θα πλαισίωναν μια τέτοια συζήτηση. Ευχαριστώ. Σαράι απόστα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Σαν Τζούλια Κίνγκ στο, στην επιστολή σας δεν αναφέρεστε καθόλου στη συνεργασία με τις φορείς της κοινωνίας των πολιτών για τις τρεις προτεραιότητες. Ε, αντιμετώπιση των τρομοκρατών, πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος. Όμως συχνά αυτοί είναι που εργάζονται στον τομέα των ε, βασικών ε, θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κύριο ρόλο στην καταπολέμηση της δροσπαστικοποίησης, την πρόληψη αυτής και της δημοκρατίας. Έχετε πρόθεση να συνεργαστείτε λοιπόν με τις φορείς κοινωνίας των πολιτών και ποια μορφή πρέπει να έχει αυτή η συνεργασία. Δεύτερον, η ομάδα σας ε, είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση όλων των μορφών της, ε, του βίου εξτρεμισμού, όπως παραδείγματος χάρη και της ε, βίας της άκρας δεξιάς. Ε, απάντηση. Θα ήθελα για κάποια στοιχεία να επιμείνω. Σε σχέση με αυτό που είπατε ε, στο τελευταίο σκέλος ερώτησης. σας, υπάρχουν, και είναι σημαντικό να το ξέρουμε, διάφορες μορφές ριζοσπαστικοποίησης. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο έναν τύπο ριζοσπαστικοποίηση. Και ε, αυτό με φέρνει στο δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσω. Ελπίζω αν εγκριθεί η υποψηφιότητά μου να μπορέσω να αντιλήσω δάγματα από την παρελθούσα μου εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας Σημαντική εμπειρία απέκτησα στην Βόρεια Ιρλανδία και εκεί αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της ρουσφαστικοποίησης. Προφανώς μια εντελώ διαφορετική μορφή της, όμως σε διάφορα βήματα της κοινότητας υπήρχε παρότρινση προς τέτοιες μορφές βίας και όπως σας είπα νωρίτερα ε, δεν μπορούσε το κράτος εκεί από ψηλά να δράσει αποτελεσματικά μόνο οι τοπικοί φορείς έχουν αυτή τη δυνατότητα. Λέω, να ενισχύσουμε στην επιστολή μου, να ενισχύσουμε την ε, απόκρισή μας στον τομέα της ασφάλειας για, ε, για το πρόβλημα της ροσπαστικοποίησης. Αυτό εννοώ. Ε, με, με, τους, με βασικούς φορείς να συνεργαστούμε. Στη Βόρεια Ιρλανδία διαπιστώσαμε ότι πολλοί εξόπιστες φωνές είναι οι πρώην κρατούμενοι. με διάφορες ομάδες Ε, καταδίκων, πρώην καταδίκων ε, συνεργαστήκαμε και υπήρξε κατάλληλη ενημέρωση και είδα πόσο αποτελεσματικό είδα. Είδα εγώ, ειδής όμως τα πρακτικά αποτελέσματα αυτή της δράσης. Και έστω και ένα νέο να εμποδίσουμε, να μην ακολουθήσει αυτό το δρόμο του ε, βίαιου εξτρεμισμού, εμένα μου αρκεί. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε επίπεδο σε μικρή κλίμακα στη Βόρεια Ιρλανδία μπορούμε να το κάνουμε και ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στους αρμοδίους φορείς. Σας ευχαριστούμε. Ερώτηση 41. Λέναρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η υποψηφιότητά σα αρχίζει σε μια ιστορική στιγμή για τι σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο και είπατε ότι δεν μπορείτε να σχολιάσετε τι διαπραγματεύσει για τον Brexit. Το σέβομαι, αλλά θα πρέπει να, σημού, να ληφθούν κάποιε αποφάσεις προσεχώ και ένα από τα πράγματα αυτά είναι η Europol. Είπατε πω πρέπει να ενισχύσουμε την Europol, να χρησιμοποιήσουμε τη νέα εντολή τη Ταυτόχρονα βλέπουμε πως η Βρετανική κυβέρνηση που σας όρισε φαίνεται πως ε, θα μείνει εκτός Europol. Πώς αξιολογείτε εσείς την αναγκαιότητα της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στη Europol και θεωρείτε πως ένα τέτοιο οπτάτ θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο το οποίο θα κάνατε ως ε, Επίτροπος για την Ένωση Ασφαλείας. Κοιτάξτε, δεν εκπροσωπώ τη Βρετανική κυβέρνηση δεν μπορώ να προκαταλάβω τις αποφάσεις της Βρετανικής κυβέρνησης αλλά θέλω να είμαι σοφής θεωρώ πως η Γεροπολή είναι ένας έξοχος οργανισμός που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και εάν τελικά όχι στο Επιτροπός θα κάνω ό,τι μπορώ για να την υπερασπιστώ και να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη εντός των πλαισίων των συνθήκων, το είπαμε αυτό, να εμπλακούν με τη πόλη. Χωρίς α, ε, κάποια διάκριση, όλα τα κράτη-μέλη. Και συγκεκριμένα για το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια πρόκληση. Πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για το εάν θα ενταχθούν ή όχι στην Europol. Αν επιλέξουν να μην το κάνουν υπάρχει πρόβλημα γιατί θα υπάρχει ένα κενό μέχρι να προσθεθεί με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου η δυνατότητα συμμετοχής μιας τρίτης χώρας. Οπότε αυτό το οποίο θα αναφέρω είναι πως είναι προς το συμφέρον όλων μας να μην υπάρξει αυτό το κενό. Καλή ερώτηση και καλή απάντηση, αν μου επιτρέπετε. Θα επανέλθω τώρα στην ουδετερότητά μου. Έχω κουραστεί, κουραστεί, συγχωρήστε μου. Λοιπόν, ερώτηση 42. Ο κύριος Λόπεζ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, υποψήφι επίτρεπε. Η ερώτηση που θέλω να θέσω αφορά την πτυχή της λογοδοσίας ε, των αναμενόμενων ε, αποτελεσμάτων που θα παρουσιάσετε. Γιατί εμείς ε, έχουμε το ρόλο να ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό έχει να κάνει καταρχήν με την επιστολή περιγραφής κατεχόντων που αφορά το χαρτοφυλακείο σας, γιατί θα πρέπει να υποστηρίξετε τον Επίτροπο Αβραμόπουλο αφενός και αφετέρου να συνεργαστείτε στενά με την Επιτροπό Γιουρόβα σε θέματα όπως η ριζοσπαστικοποίηση και η ανταλλαγή πληροφοριών. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με την ισορροπία που θα πρέπει να βρείτε μεταξύ των καθηκόντων σας ε, απέναντι σε πολλούς επιτρόπους πόσο ανεξάρτητος ε, προβλέπετε ότι θα είστε στην επιτέλεση του καθηκόντων σας και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο θα επισκευαστεί συγκεκριμένα από τον Επίτροπο Ευρωμόπουλο και μείνετε εδώ παρακαλώ γιατί έχετε ξεπεράσει το χρόνο. 1,5 λεπτό έχετε μιλήσει. Ένα τελευταίο σημείο για την αρχή τη λογοδοσία απέναντι σε αυτήν την Επιτροπή, ενώπιον αυτές τι Επιτροπές, Καθώ στην επιστολή περιγραφή καθηκόντων σα λέγεται ότι αυτά τα καθήκοντά σου που αφορούν την ασφάλεια δεν θα επιτελούνται αποκλειστικά από τον Επιτρόπο Αβραμόπουλο. Ευχαριστώ. Καλώ ορίζω τι ερωτήσει σας, γιατί μου δίνουν και πάλι την ευκαιρία να εξηγήσω, όπως έκανα και σε κάποιες από τις γραπτές μου απαντήσεις, πώς ελπίζω ότι θα λειτουργήσει όλο αυτό. Δεν έχω πρόβλημα με αυτή τη συζήτηση που τίθεται περί της σκίασης κτλ. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι συνάδει με τη σημασία αυτού του ρόλου. Εδώ αυτός ο ρόλος δεν είναι ε, δεύτερος ρόλος, ούτε είναι μερική απασχόληση, αλλά εγώ, βάσει και του δικού μου πολιτικού πολιτισμού, θα θέλω να συνεργαστώ στενά με τους υπόλοιπους επιτρόπους και ιδίω με τον Επιτρόπο Αβραμόπουλο, αλλά και όχι μόνο, με μια σειρά συναδέλφων επιτρόπων ε, για μια σειρά θεμάτων που έχουμε συζητήσει απόψε. Γιατί μαζί νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το θεματολόγιο σε ό,τι αφορά τώρα τη λογοδοσία απέναντί σα, όπω είπα από την αρχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που λογοδοτώ σε εσά ε, και θα λογοδοτήσω σε εσά οποτεδήποτε θέλετε να μου μιλήσετε. Και φυσικά θα λογοδοτώ απέναντί σας για τη διάσταση ασφαλείας οποιοδήποτε, οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα. Εσείς θα κρίνετε, αλλά νομίζω ότι εν τέλει θα έχετε μία σημαντική αύξηση της λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον αυτού του Κοινοβουλίου και υπό αυτό το πνεύμα θέλω να προσεγγίσω το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Περνάμε στην ερώτηση 43. Η κυρία Μαρία Καμπριέλ για τη ερώτηση το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κίνγκ, Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων στη Βουλγαρία. Αυτό αφορά και την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το εξής. Η Βουλγαρία ε, δεν έχει πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων ΣΥΣ, ενώ δίνει για χρόνια πληροφορίες και αυτό μπορεί να θέτει ενδυνάμει κίνδυνο στην ασφάλεια της Ένωσης. Τι, θα, τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε η χώρα που πληρεί τα τεχνικά κριτήρια για την ένταξη στις ε, ΣΕΝΓΕΝ να μπορεί να συνεισφέρει και να έχει πρόσβαση στην πραγματική ανταλλαγή δεδομένων, όπως είπατε. Και ερώτηση υπαριθμών 2. Ανησυχείτε σας ανησυχεί το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, δώσει ευρωπαϊκά διαβατήρια σε ανθρώπου από τρίτε χώρες και τρίτον εσείς ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε την τρομοκρατία στη Μεσόγειο η ασφάλεια της Μεσογείου σημαίνει και ασφάλεια στην Ευρώπη σας ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ για την κατάσταση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το συζητήσαμε αυτό και λίγο νωρίτερα. Πραγματικά κατανοώ τις ερωτήσεις που μου θέτετε. Η Βουλγαρία μπορεί να δει τις καταχωρήσεις για τις απορρίψεις, για τις αρνήσεις, αλλά δεν μπορεί να λάβει δράση από αυτών. Και νομίζω ότι είναι μια πραγματική ερώτηση. Είναι προ το συλλογικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι τέτοιο νομικά. Είναι σαφή η κατάσταση. Έρονται οι περιορισμοί όταν τα κράτη-μέλη τη Σέγγεν το αποφασίσουν. όμω πολιτικά κατανοώ την ερώτηση και νομίζω ότι είναι νόμιμο να ρωτάτε αν στι σημερινέ συνδικέ δεδομένε τη απειλή που αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά κατά τέτοιο εξυπηρετεί το συλλογικό συμφέρον. Τώρα, για την ερώτηση των διαβατηρίων, περί των διαβατηρίων. Και βέβαια και το θέμα της υπηκότητας. Το θίξαμε αυτό. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά όταν δίνει κάποιος υπηκότητα ενό κράτου μέλου, ουσιαστικά δίνει υπηκότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι επομένω τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουν κατά νου το συλλογικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν λαμβάνουν αυτή την απόφαση και φυσικά και τα θέματα ασφαλείας. Όταν ε, λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τους επισημαίνουμε να είναι σόφρονα. Σας ευχαριστούμε και τελική ερώτηση 44 από την κυρία Γκόμες από τους Σοσιαλιστές. Julian King. Ε, υπάρχουν αποδείξει ότι οι τρομοκρατικέ οργανώσει χρηματοδοτούν τι επιχειρήσει του μέσω οργανωμένη εγκληματικότητα. Μιλήσαμε για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων και απαντήσατε. Όμω θεωρείτε ότι υπάρχουν κενά το ελληνικό σύστημα για την αντιμετώπιση αυτού του συστήματο χρηματοδότηση, διότι η νομιμοποίηση εσόδων γίνεται μέσα στις χώρες ΟΠΕΚ και σε συστήματα συνεργασία που, ε, ε, στα οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκές τράπεζες, μεσητικά γραφεία, σύμβουλοι, consultants, ε, χρησιμοποιούν φορολογικού παραδείσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού και υπάρχει το, η κοινή ανησυχία με αυτά τα συστήματα των χρυσών ε, θεωρήσεων που ε, τα κράτη-μέλη προσφέρουν. νομίζω ότι αναφερθήκατε έτσι φευγαλέα σε αυτό στην τελευταία σας ερώτηση. Έχετε κάποια πρόθεση να διασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση, διότι επανερχόμαστε σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας ε, για τη δράση που θέλω να αναλάβω συγκεκριμένα. Ε, να διακόψουμε ε, την ε, πρόσβαση των τρομοκρατών στη χρηματοδότηση. Μιλήσαμε για την κατάσχεση πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για την, τις πηγές χρηματοδότησης και ε, επίσης ενίσχυση των ε, μέσων που έχουμε για την καταστολή της τρομοκρατίας και εξετάζω σοβαρά το ενδεχόμενο ε, να κάνουμε κάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι πολύ αποτελεσματική η συνεργασία μέχρι στιγμής με τη ΣΥΠΑ, παραδείγματος χάρη. Ε, πολλά μπορούμε να κάνουμε, πολλά θέλω να κάνουμε και θέλουμε να ενισχύσουμε σίγουρα τη διεθνή συνεργασία για την καταστολή της διαφθοράς, της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και της κατάχρησης κάποιων οχημάτων χρηματοδοτικών οχημάτων για την χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Μετά τις εργασίες της ομάδα G7 και G20 για το θέμα αυτό και σας παραπέμπω και σε αυτά που έκανε ε, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κάμερον, την άνοιξη του 2016 για την ενίσχυση της διεθνούς ε, συνεργασίας ε, σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Μπορούμε να δώσουμε συνέχεια και όταν, ε, άμα μας δοθεί η ευκαιρία και αν σημειωθεί πρόοδος στα επόμενα χρόνια, με χαρά θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση από... και ε, ε με ράντεβε τελευταία ερώτηση από πλευρός του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλημμυρίσει μετανάστες και κάποιοι από αυτούς ε, δυστυχώς ε, διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα παράνομα. Ε, είναι αδύνατον για κάποιους από τους ανθρώπους να ελέγξουμε ποιοι είναι για να δούμε αν ανήκουν σε τρομοκρατική οργάνωση. Τι θα κάνετε εσείς ως αρμόδιος επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια για να μην υπάρχει ο κίνδυνος ρίζος και τρομοκρατικών ε, επιθέσεων από μετανάστες που φτάνουν στην Ευρώπη, ειδικά από αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Uh, thank you. Um... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν νομίζω πολλές πιθανές αιτίε ε, ριζοσπαστικοποίησης, θεωρώ. Και νομίζω μια αίσθηση απομόνωσης και αδικές μπορεί να παίξει το ρόλο της. Η αντίδραση νομίζω πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη όπως είπαμε Να αντιμετωπίσουμε δηλαδή την προπαγάνδα μίσους, την αντιμετώπιση της ρίσοσπαστικοποίησης στα σχολεία, την αντιστροφή της στις φυλακές και βεβαίως να είμαστε αποτελεσματικοί στις πολιτικές ένταξεις. Είναι κάτι το διαφορετικό από την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίηση αλλά πρέπει, αν βοηθάει, να το κάνουμε και αυτό. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης ε, για την ε, ένταξη, την ενσωμάτωση, το οποίο θέλω να συζητήσω με τους συναδέλφους, γιατί και εδώ πέρα απαιτείται ομαδική προσπάθεια για να σημειώσουμε πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έμειναν για ολόκληρη την συνεδρίαση και ευχαριστώ ιδιαίτερα έμειναν όπως ήρθαν από την αρχή και έμειναν. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σα. Περνάμε τώρα στην ε, τελική μίληση του κυρίου Κίνγκ, του υποψηφίου Επιτρόπου για 5 λεπτά. Σας παρακαλώ να μείνετε και μετά από αυτή τη σύνδεση. Και εγώ θέλω να φύγω, να μην εξαφανιστείτε. Το είπα δυνατά, το είπα. Ε. Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για το τι θα, πώς θα αποφασίσουμε δημοκρατικά για τον υποψήφιο επίτροπο. Παραμείνετε λοιπόν για λίγα λεπτά. Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον υποψήφιο επιτροπό να κάνει μια δήλωση μέχρι πέντε λεπτά, αν θέλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές για τις ερωτήσεις σας και για το ότι με ακούσατε και για την υπομονή που επιδείξατε. Ας δούμε αν θα περιοριστώ αυτή τη φορά χρονικά, αν θα μπορέσω να νικήσω το ρολόι. Νομίζω πως είναι προφανές από τις τελευταίες ώρες, τις συζητήσεις μας, πως υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και αν τελικά οριστό ε, επίτροπος. Θέλω να αναλάβω καθήκοντα το συντομότερο δυνατόν. Όπως είπα στην αρχή, θεωρώ εαυτόν πλήρως υπόλογο σε εσάς και θέλω να αναπτύξουμε στενές σχέσεις. Οι συμπολίτε μας ε, δικαιολογημένα ανησυχούν για την αύξηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και περιμένουν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαντήσουμε. Η απάντησή μας πρέπει να είναι συλλογική, συντονισμένη και συνολική. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και τη δουλειά που γίνεται σε διάφορα μέτωπα να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και να ενισχύσουμε την άμυνά μας με τρόπο ο οποίος θα σέβεται τις αξίες μας και τα θεμελιώδη δικαιώματα συμφωνήσετε με τον διορισμό μου θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να συνεργαστούμε, για να κάνουμε την Ευρώπη ασφαλέστερη. Θα πρέπει λοιπόν ο στόχο να έχουμε την ελευθερία και ασφάλεια όλων των ανθρώπων που ζουν και ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με έναν τρόπο ο οποίος θα βασίζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες. Και έτσι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προλάβουμε την ριζοσπαστικοποίηση και το οργανωμένο έγκλημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. So in answering my plea, colleagues, you're not running. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ που δεν τρέξατε να φύγετε. Ε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο για να γίνετε αρεστός εδώ πέρα. Δεν εξαντλήσατε το χρόνο που σας ε, αναλογούσε. Ε, συνάδελφοι, οι συντονιστές θα συσκεφτούν αύριο στις 13 Σεπτεμβρίου στις 9 Εξ ονόματός σας θα αποφασίσουν οι συντονιστές ε, αν ε, πληρεί ο επιψήφιος τα πρότυπα που επιθυμούμε για να μπορέσει να επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά του. Αύριο είναι λοιπόν η σύσκεψη και μετά θα ενημερώσω τι πολιτικές ομάδες. Αν δεν υπάρχουν ενστάσει, ε, θα μάθετε μετά την κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση των συντονιστών τι ε, Σας ευχαριστούμε που Ήσασταν εδώ, όχι μόνο τα μέλη της ΛΥΜΠΕ, συνάδελφοι από την ΑΦΕΤ και άλλοι συνάδελφοι από άλλες επιτροπές που ήρθαν και δεν ε, πήραν το λόγο. Τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ τα ευχαριστώ όλους ιδιαίτερως. Ήσασταν τόσο μεθοδικοί στη δουλειά σας ε, και σχολαστικοί και σας ευχαριστούμε ε, σε Τζουλιαν Κίνγκ. Κατά πάσα πιθανότητα δεν χρειαστεί να κάνετε κάτι άλλο αντίστοιχο στην σταδιοδρομία σας εφ' Είναι πάρα πολύ σημαντική η Ένωση για την Ασφάλεια και αν δείτε στο Twitter φαίνονται όλα πολύ πιο σανροπαστικά από ό,τι ήταν πραγματικά στην αίθουσα. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ε, χαρτοφυλάκιό σα. Εμείς ε, πραγματικά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ε, σε όλα αυτά τα ζητήματα και προσβλέπουμε ενδεχομένως μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστούμε.